Hello, good afternoon. Please. Καλησπέρα, καθίστε παρακαλώ. Good afternoon to everybody. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο εργαστήριο που διοργανώνει η Επιτροπή Αναφορών. Καλέσαμε για το εργαστήριο αυτό κάποιους εμπειρογνώμονες. Δύο από αυτούς κάθονται δίπλα μου και αναφέρονται στον πιο σχετικών αναφορών για το σχιστοδυσικό αέριο, φυσικό αέριο. Καλέσαμε δύο συγγητές της Ήτρε και της Ένβη που συντάσσουν εκθέσεις, την κυρία Τζαβέλα και τον κύριο Σόνικ. Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε τις πρώτες υποχωρήσεις το 2011 και οι παλαιότερες είχαν τεθεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2012. Κάποιες αναφορές είναι αρκετά γενικές, αναφέρουν γενικές ανησυχίες για περιβαλλοντικές πτυχές και τι αντίκτυπο έχει στο έδαφος ε, η μέθοδος εξόριξης ε, αυτών των ειδών αερίων από σχιστόλιθο ε, οι βασικέ χώρε που ασχολούνται το θέμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η εξόριξη διαφόρων ειδών αερίου μη τυπικών είναι σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ε, οι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το θέμα και σε κάποιες χώρες και περιοχές και περιφέρειες ε, γίνονται μαζικέ διαμαρτυρίε. Γαλλία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποφάσισαν να επιβάλλουν ένα μορατόριο όσον αφορά εξαγωγή συστολιστικού αερίου που αναφέρεται σε υδρορογμάτωση. Μέχρι ότου έχουν εξελιχθεί περισσότερες τεχνολογίες. Κάποιοι αναφέροντες πιστεύουν ότι το παρόν νομικό πλαίσιο που ισχύει για την υδρορογμάτωση είναι ανεπαρκές και υπάρχουν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Ακριβείς ερωτήσεις έχουν τεθεί και έχουν υποβληθεί και κάποιες προτάσεις σχετικά με το θέμα. Η αναθεώρηση των κατοφλίων που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο παράρτημα όσον αφορά τις εξολογήσεις αντιχτύπου για το περιβάλλον και σχετικές οδηγίες που διέπουν η υδρολυτική, ε, υδρολυτική, επιφανειακή υδρολυτική εξόριξη ίσως επηρεάζει τα επιφανειακά ύδατα και δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για τα ύδατα. Και η χρήση χημικών ουσιών για την υδροφραγμάτωση ε, είναι κάτι που απασχολεί και ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τι δραστηριότητε. Κάποιοι αναφέροντε λένε ότι η προσπάθεια ανακάλυψη του αερίου και ο τρόπο εξόριξη ε, θα πρέπει να οδηγήσει τελικά σε μείωση της χρήσης ε, ορυκτών καυσίμων και την μείωση εκπομπών. Ε, έχουν εδώ συσταθεί πολλές, πολλά εργαστήρια, πολλές ακροάσεις έγιναν, πολλές εκθέσεις έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές επί του θέματος. Να επιθυμίσω την ακρόαση που διοργανώθηκε την Επιτροπή Ήτρε, όσον αφορά την προοπτική για την χρήση συστολιθικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Οκτωβρίου του 2011 και το εργαστήριο που διοργανώθηκε την Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει η εξαγωγή συστολιθικού αερίου και πετρελαίου ε, στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία το Φεβράριο του 2012 το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Ολομελίας του Οκτωβριού θα υιοθετήσει δύο σημαντικές εκθέσεις. Η μία από την Επιτροπή Βιομηχανίας, η έκθεση για την βιομηχανική ενέργεια και άλλες πτυχές ε, του συστολιθικού αερίου και πετρελαίου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Νίκη Τζαβέλα και έχουμε και άλλη μια έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την έκθεση για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εξόριξης συστολιθικού αερίου και πετρελαίου και των σχετικών δραστηριοτήτων που η είναι ο κ. Μπούκος Λαυσόνικ. Οι δύο εισηγητές προσεκλήθησαν, όπως σας είπα και στην αρχή, να παραστούν στο εργαστήριό μας και να μοιραστούν μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις που διαθέτουν στον τομέα. Δεν γνωρίζω αν θα είναι παρόντες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε τρεις μελέτες σχετικά τα μη συμβατά ορυκτά καύσιμα, κάτι που ανέλαβαν εξωτερική συμβουλή. Αυτές οι μελέτες εξετάζουν αντίστοιχα τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των καυσίμων όσον αφορά τις ενεργειακές αγορές, τις ενδεχόμενες ε, συνέπειες που θα έχει η παραγωγή συστολιστικού αερίου στο περιβάλλον και κατά πόσο οι όλε διαδικασίε αυτέ έχουν συνέπειε στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το εργαστήριο ε, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Βασικό σκοπό είναι να ανταποκριθεί στα ερωτήματα των αναφερόντων και ταυτόχρονα να δώσει στα μέλη ε, πολύτιμε ιδέε για τι μελλοντικέ εργασίε όσον αφορά την διερεύνηση για σχιστολιθικό αέριο και την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου. Ε, θα ξεκινήσουμε Μου λέγουν ότι κατέφθασε ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Ματίας Αλτμαν, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τη μελέτη για τον αντίκτυπο που έχει εξόριξη ισχύ στο λιθικό αερίο στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ενημερωμένης μελέτης. Μπορείτε παρακαλώ να βάλετε 100% την εικόνα στην οθόνη. Πρόκειται για ενημέρωση. Βασίζεται λοιπόν στη μελέτη που κάναμε πριν από ένα έτος ακριβώς για την Επιτροπή Περιβάλλοντος Κυρίως ασχοληθήκαμε με τα νέα θέματα που προέκυψαν μετά την προηγούμενη μελέτη, όπου δηλαδή υπήρξε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την επιστημονική γνώση. Το αναφέρουμε σε αυτή τη μελέτη που ε, υπάρχει και έντυπα και θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονικός. Υπάρχουν έξι τμήματα. Δεν θα διαβάσω όλα όσα λέει η κάθε διαφάνεια. Θα ασχοληθώ με τα κυριότερα και ε, μετά μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες. Τα περισσότερα που αναφέρω εδώ βασίζονται σε πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες, τρεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήδη ανέφερε η κυρία Ματσόνη, οι άλλες είναι κυρίως μελέτες που παρήγγειλαν γερμανικές αρχές, εθνικές και περιφερειακές. Τρεις χιλιάδες σελίδες συνολικά ε, επιστημονικού κειμένου. Νομίζω ότι είναι ήδη μια τεκμηριωμένη βάση συζήτησης. Όμως υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά Αυτό είναι λυπηρό γιατί στι ΗΠΑ έχουμε τόσο μεγάλη πείρα. Υπάρχει σημαντική βιομηχανική χρήση. Οπότε τα στοιχεία θα μπορούσαμε να τα έχουμε για να τα αναλύσουμε. Μία μελέτη που ήδη αναφέρθηκε, που την παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνει μια πρώτη προσπάθεια να κάνει μια συνολική αποτίμηση του κινδύνου για μη συμβατικές μεθόδους ε, εξόρυξης φυσικού αερίου, συγκεκριμένα υδρορογμάτωση. Βλέπετε εδώ τις δύο κολόνες, βλέπετε αναέργο και αθρηστικό αποτέλεσμα των μη συμβατικών μορφών εξόρυξης. Βλέπετε ότι γενικά η μη συμβατική εξόρυξη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει συσσόρευση πολλών μεμονωμένων ε, πηγαδιών. Φρε, φρεατίων. Μπορεί σε ένα χωράφι να έχουμε χίλια φρεάτια, ας πούμε. Στη μεσαία στήλη εδώ βλέπετε τους κινδύνους που ποιοτικά θεωρούνται μέσου επίπεδου, άλλοι υψηλού ή άλλοι χαμηλού επίπεδου. Αλλά αν δείτε αθρηστικά το αποτέλεσμα, θα διαπιστώσετε ότι αθρηστικά είναι υψηλού επίπεδου κινδύνου. Δεν μπορώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για όλα αυτά. Μερικά στοιχεία θα εξετάσω αναλυτικότερα στις επόμενες ε, σελίδες. Παράδειγμα, εκκλήσεις αερίων στον αέρα. Όπως βλέπετε, ένα φρεάτιο δεν είναι τόσο μεγάλος κίνδυνος, αλλά το θρηστικό αποτέλεσμα βεβαίως αυξάνει τον κίνδυνο. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε τις διάφορες φάσεις της εκμετάλλευσης. Από την ταυτοποίηση του χώρου, προετοιμασία του φρεατίου, μέχρι τέλους εγκατάλειψη του φρεατίου και την ε, αντιμετώπιση μετά την εγκατάλειψη της παραγωγής. Γεωλογικές πλευρές τώρα, πολύ σημαντικές. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ε, για το τι γίνεται μεταξύ 100 και 2.000 μέτρων. Διότι εδώ αυτό το στρώμα είναι απλώς μια προστατευτική ζώνη ανάμεσα στο, στους υδρογονάνθρακες και τα υπόγεια ύδατα που είναι παραπάνω. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή, η, αυτό το στρώμα ως ε, φράγμα οι γεωλογικές ε, διαδρομές ε, θα εμφανιστούν ε, στην επόμενη σελίδα. Εκτός από την θεωρητική γεωλογική ανάλυση και την ανάλυση που βασίζεται στις διερευνητικές γεωτρήσεις, μας ενδιαφέρει να ελέγχουμε την ποιότητα του ποσίμου ύδατος για να δούμε όσο δυνατόν νωρίτερα τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα αυτών των μη συμβατικών μορφών εξόριξης. Ας δούμε τις διάφορες διαδικασίες πώς ε, διεξάγονται στο επέδαφος. Βλέπουμε ότι πολύ βαθιά γίνεται η υδροορογμάτωση και περνάει από τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν είναι πάντα παρόν υδροφόρος ορίζον, αλλά μπορεί να υπάρχουν γεωλογικά ασφάλματα. Οπότε θα μεταφερθούν χημικές ουσίες από το βαθύτερο στρώμα του αερίου στα ύδατα. Πρέπει λοιπόν αυτές οι γεωτρήσεις να γίνονται εκεί που δεν υπάρχουν γεωλογικά σφάλματα ή ρήγματα και τα παλιά εγκαταλειδημένα φρεάτια μπορεί επίσης να παίξουν το ρόλο διόδου από τα πιο βαθιά στρώματα στα παραπάνω. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ρινανία Ερνανία-Βεστφαλία, όπου υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτή τη δραστηριότητα. Έχει πολλές γεωτρήσεις, 60.000 παλιές γεωτρήσεις, ορισμένες ε, εδώ και δεκαετίες. Για ορισμένες ούτε ξέρουμε πού ακριβώς είναι. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η τρίτη δυνατή δηλαδή διαδρομή είναι μέσω το αδια... μέσω του αδιαπέρατου πετρώματος αλλά παρά το ότι λέγεται αδιαπέρατο, μπορεί να περάσουν ε, κάποια υγρά. Ε, και βεβαίως και η ίδια η γεώτρηση διαρριγνύει την ε, ακαιρεότητα των στρωμάτων και μπορεί να χρησιμεύσει ως δίωδος. ο κατακαιρματισμός είναι ένα θέμα, μπορεί να παίξει ρόλο. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παρατηρούμε κατά πόσο παραμένει μετά την υδρορογμάτωση επαρκώς άθικτο το πέτρωμα γιατί μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Θα πρέπει να μελετάμε πάντα αν υπάρχουν ρήγματα στα διάφορα γεωλογικά στρώματα. Αυτό δεν μπορεί να αναλυθεί γενικώ. Πρέπει να αναλύεται κατά περίπτωση. Μέσω του αδιάρρηκτου πετρώματος περνάει βέβαια το αέριο. Έχει γίνει μια μελέτη και θεωρούν ότι σε 30 χρόνια είναι περιορισμένη αυτή η μετάδοση. Θεωρούν ότι μπορεί να, πάει, ε, να, να προχωρήσει το αέριο 50 εκατόμετρα οι διάφορες ουσίες. 30 χρόνια λοιπόν είναι το πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε. Οπότε για πάνω από 30 χρόνια δεν έχουμε στοιχεία. Αυτό το αναγνωρίζουν όλες οι επιστημονικές μελέτες. Γιατί αναφέρθηκα στα 50 εκατό μέτρα. Αν επιχειρήσουμε να βρούμε λοιπόν ε, πόσο μακριά από τον υδροφόρο ορίζοντα πρέπει να γίνει η υδρορογμάτωση, οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι χρειάζονται 600 συν 300 μέτρα για τα άνω στρώματα που δεν θεωρούνται αδιαπέραστα γιατί δεν είναι τόσο πυκνά όπως τα παρακάτω στρώματα. Θεωρούν λοιπόν οι επιστήμονες ότι αυτή η γεώτρηση πρέπει να είναι τουλάχιστον χίλια μέτρα βαθιά. Και αν υπάρχουν ε, βαθύτερα υδροφόροι ορίζοντες που χρησιμοποιούνται, το πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 600 μέτρων καθέτος ως ε, περιθώριο ασφαλείας, ως ζώνη ασφαλείας. Λοιπόν, ποιε ποιες χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται για την υδρορογμάτωση, είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μία από τις δύο βασικές αιτίες ενδεχόμενης ε, μόλυνσης. Αναμειγνύουμε λοιπόν αυτές τις ουσίες με νερό και με κάποιο προθετικό όπως άμμο και αυτά τοποθετούνται μέσα, ε, πιέζονται μέσα στην ε, γεώτρηση. Προωθούνται λοιπόν όλα αυτά με στη γεώτρηση και έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ διαφορετικές ουσίες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική. 150 χημικές ουσίες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στη Γερμανία. Έχουν γίνει περίπου 300 υδρορογματώσεις. Μια πολύ αναλυτική επιστημονική μελέτη των χημικών ουσιών έχει καταλήξει σωσμένα συμπεράσματα. Πρώτον, οι μισές περίπου, περίπου χημικές αυτές ουσίες μπορούν να αναγνωριστούν μέσω των πληροφοριών που μας δίνουν οι ε, εταιρείες που εκμεταλλεύονται το κοίτασμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τις πληροφορίες μας έδωσε η Exxon Mobile. Για τις άλλες ουσίες έγινε επιστημονική προσπάθεια να τις καθορίσουμε να τι αναγνωρίσουμε και τις μισές περίπου δεν καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε, κάτι που είναι δύσκολο βέβαια, κάτι που δεν μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο τοξικές είναι. Πόσο τοξικές είναι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι να συσχετίσουμε τις συγκεντρώσεις χημικών στο υδρορογματικό υγρό με το αποτέλεσμά τους. Δηλαδή, Πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει. Έχουμε την λεγόμενη έννοια της ε, δραστικής συγκέντρωσης. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δραστική μια συγκέντρωση όταν, για παράδειγμα, δολοφονεί 50% των ζώων με το οποίο έρχεται σε επαφή. Ή μια άλλη ε, παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι η μια αλλη παραμετρο που λαμβανεται υποψη ειναι η συγκεντρωση που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτές οι αναλύσεις κάναμε για όλες τις χημικές ουσίες που καταφέραμε να αναγνωρίσουμε. Εδώ βλέπετε ένα πίνακα που ε, συγκρίνει μερικές από τις ουσίες που ε, αναγνώρισαν αυτές οι μελέτες. Βλέπετε λοιπόν ότι οι συγκεντρώσεις που θεωρούν ε, επικίνδυνες οι δύο μελέτες απέχουν πολύ. Ε, έχουμε διαφορές στις τάξεις του 10, 100 έως και 10.000. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ποια συγκέντρωση μας ενδιαφέρει. Βεβαίως, μια συγκέντρωση που δεν έχει καθόλου αποτέλεσμα πρέπει να ορίζεται με βάση ένα πολύ μικρό αποτέλεσμα θανάτων στα ζώα κτλ. Αλλά βλέπετε δύο παραδείγματα στα κόκκινα παραλληλόγραμμα που αποδεικνύουν ότι και για τις αναλύσεις αυτές υπάρχουν διαφορές. Για μένα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για να δούμε ποιες συγκεντρώσεις έχουν ε, βλαβερά αποτελέσματα και ποιες όχι. Άλλο σημαντικό θέμα. Τι να κάνουμε με το μολυσμένο νερό. Τι είναι μολυσμένο νερό στα πλαίσια της συζήτησης αυτής. είναι αποτέλεσμα του υδρορογματικού υγρού που προωθείται. Αλλά και στα παραπάνω στρώματα υπάρχει νερό που και αυτό μπορεί να περιέχει υψηλό ποσοστό τοξικών και επικινδύνων ουσιών. Τα είδατε λοιπόν αυτά και αυτά ανεβαίνουν προς τα πάνω μέσω της υδρορογμάτωσης. Βλέπετε διάφορες συγκεντρώσεις σε αυτό το διάγραμμα το πιο σκοτεινό κομμάτι είναι νερό που ήδη υπήρχε μέσα στη γη ενώ το πάνω κομμάτι προκύπτει από το, από το υδρορογματικό υγρό. Οπότε, κατά την υδρορογμάτωση, το υγρό που ανεβαίνει πάλι μέσα από το φρεάτιο συναντάται με το νερό που υπάρχει παραπάνω. Δηλαδή αν το υγρό αυτό ακόμη και αν δεν έχει καθόλου χημικές ουσίες, πρέπει να δούμε πώς θα επεξεργαστούμε αυτό το νερό που ανεβαίνει από τα φρεάτια, γιατί μπορεί παρόλα αυτά να είναι επικίνδυνο. Επίσης ένα τμήμα του υδρορογματικού υγρού μένει μέσα στη γη, δεν θα ανέβει μέσω της διαδικασίας της αναρροής. Έχουμε μια σειρά από δυνατότητες ε, αντιμετώπισης του υγρού αναρροής αυτού. Στη Γερμανία γενικά το επανεγχύουν σε ένα άλλο σημείο, σε βαθιούς, βαθιούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Αυτή είναι η λεγόμενη γεωλογική ενταφίαση. Επίσης μπορεί να ανακυκλωθεί να χρησιμοποιηθεί το νερό για υδρογμάτωση περαιτέρω, αλλού. Ή για άλλου ε, σκοπούς. Αυτό γίνεται εν μέρει στις ΗΠΑ. Όπου αυτό το νερό χρησιμοποιείται για ενισχυμένη ε, διαδικασία αναλαβής πετρελαίου. Αυτός ο πίνακας είναι κάπως περίπλοκος. Εδώ σας, σας βάζω αυτό το πίνακα για να δείτε πώς αντιμετωπίζετε τα διάφορα στοιχεία που είναι στο υγρό αναρροής. Υπάρχει ό,τι θέλετε μέσα σε αυτό το υγρό αναρροής που είναι στην ουσία απόβλητα. Άρα θα χρειαστούν διάφορες, διαφορετικές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσετε αυτό το νερό που επιστρέφει, που ανεβαίνει πάλι πίσω. Οπότε χρειάζεται να δαπανίσουμε μεγάλα ποσοστά ενέργειας που βέβαια είναι αντιφατικό με το στόχο μας. Το πόρισμα μιας γερμανικής μελέτης γι' αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά προχωρημένη γνώση ούτε τεχνολογία για την αντιμετώπιση αυτού του υγρού που ανεβαίνει που θα επέτρεπε μετά να το χύσουμε σε έναν υδροφόρο, σε μια υδροφόρα ροή. Δηλαδή δεν μπορούμε να το κατεργαστούμε και μετά να το ρίξουμε σε ένα ποτάμι. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες. Επίσης καταλήγει η μελέτη αυτή ότι οι πρώτες ε, τεχνολογίες κατεργασίας του υγρού αυτού που χρησιμοποιήθηκαν στις ΗΠΑ δεν συμμορφούνται με τις διατάξεις ε, των νόμων προστασίας στη Γερμανία. Άρα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Τώρα, ποιος είναι ο απολογισμός από πλευράς ε, αερίου θερμοκηπίου. Πριν από ένα χρόνο κάνω αυτή την ανάλυση και είχαμε πολύ υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω της μη συμβατικής εξόρυξης φυσικού αερίου. Αυτό οφείλεται στις ε, εκπομπές μεθανίου από αυτό το υγρό που ξανανεβαίνει. Δεν περιέχει λοιπόν αυτό το υγρό μόνο ε, επικίνδυνες ουσίες, αλλά και διαλελειμμένο μεθάνιο. Αυτό που θέλουμε να βγάλουμε από τα κάτω στρώματα. Εάν λοιπόν κατόπιν εξαερωθεί αυτό το μεθάνιο, έχουμε πολύ ψηλές εκπομπές ε, αεριοθερμοκηπίου. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες πρακτικές θα αξιοποιήσουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. χαμηλά το συγκρίνουμε με το ανανεώσιμο ε, μεθάνιο που προκύπτει από το βιοαέριο για παράδειγμα ή από άλλες ε, μορφές. Εδώ είναι πολύ χαμηλές εκπομπές. Μετά βλέπετε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιέχεται σε μία μελέτη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες δημοσιεύτηκε που μας δίνει αρκετά χαμηλά στοιχεία για την υπόθεση βάσης. Α, με συγχωρείτε. Α, για το Ρωμανό Βασίλειο είναι το συμβατικό φυσικό αέριο. Το, η φάση τη πρώτη καύση είναι το γαλάζιο και η φάση καύση είναι το σκούρο μπλε. Αν το συγκρίνουμε με την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, έχουμε πολύ περισσότερο θαλασσί. Δηλαδή, η μεταφορά μέσω αγωγών από τη Ρωσία αγωγών μήκους 7.000 χιλιόμετρων προκαλεί σημαντικές ε, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αν δείτε παραπάνω το μη συμβατικό φυσικό αέριο, είναι η περίπτωση Altman που λάβουμε υπόψη πέρυσι, η παραπάνω είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μία βέλτιστη και μία χείριστη περίπτωση. Είναι και δύο χειρότερες από το συμβατικό φυσικό αέριο στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά καλύτερες από το εισαγόμενο από τη Ρωσία. Αν πάρουμε την ε, βασική υπόθεση που θέλουμε να αναλύσουμε, Υπάρχει και διοξείδιο του άνθρακα σε αυτό το αέριο που βγάζουμε από τη γη. Αν το ανεβάσουμε στην επιφάνεια, διαχωρίζεται και εξαερούται. Εξαρτάται λοιπόν πάρα πολύ από το περιεχόμενο διοξιδίου του άνθρακα, του φυσικού αερίου που εξάγουμε. Πήραμε την ε, βέλτιστη περίπτωση τη ε, μελέτη του αερίου και το εφαρμόσαμε σε ένα φυσικό αέριο που περιέχει 30% διοξείδιο του άνθρακα. Που είναι η περίπτωση σε ένα σημαντικό πεδίο σχιστολτικού αερίου στις ΗΠΑ. Είναι πραγματικά χείριστη περίπτωση. Αποδεικνύει ότι είναι ουσιαστικά χειρότερη από το συμβατικό αέριο που εισάγεται από τη Ρωσία, αλλά καλύτερο από καύση άνθρακα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Στη διάθεσή σα για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι όλες οι διαφάνειες του PowerPoint είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματο και όλες οι ομιλίες θα είναι online διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και δημοσιευθούν από το τμήμα πολιτικής σε βιβλία, σε μικρό βιβλιαράκι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αναστασίο και σας παρακαλώ αν έχει την καλοσύνη να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα του χρόνου ομιλίας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου πεθύνατε. Μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να μιλήσω σε τέτοιο δικαιωμένο κοινό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσω με την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις ενεργειακές πηγές πριν από 40 χρόνια. Ε, θέλαμε να βρούμε έναν τρίτο προμηθέα Δηλαδή να βρούμε μια εναλλακτική λύση όσον αφορά τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όσον αφορά τις εξαντλούμενες πηγές ενέργειας και τα αποθέματα, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ε, αυτό το ερώτημα που θέτουμε είναι το εξής. Τι χρησιμοποιούμε για να αντικαταστήσουμε τις συμβατικές πηγές ενέργειας, συμβατικές πρώτες ύλες. Ποιες μελλοντικές πηγές θα χρησιμοποιήσουμε θα αναφερθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι κρισίμου σημασίας. Γεωλογικός πώς πρόκειται περί αποθεμάτων που εμπεριέχουν πετρέλαιο. Συνεπάγεται ότι έχουμε ένα επίπεδο μία λεκάνη που δέχεται ουσιαστικά τη που περνάνε από την πηγή. Έχουμε επίσης μία παγίδα αν θέλετε, μία λεκάνη ε, απορροής και το αέριο το οποίο διαμορφώνεται στο μητρικό πέτρωμα είναι ε, φυσικό αέριο που είναι μια συμβατική πηγή ενέργειας που λαμβάνουμε υπόψη. Μιλάμε για μη συμβατικές πηγές και το σχιστολιθικό αέριο πιο συγκεκριμένα πρέπει να δεχτούμε ότι τα παλιά γεωλογικά μορφώματα, οι παλιοί βράχοι έχουν γίνει αποθέματα ουσιαστικά, αποθεματικοί χώροι. Και πώς μπορούμε να πάρουμε το αέριο από εκεί για να το χρησιμοποιήσουμε όπως θα χρησιμοποιούσαμε ένα συμβατικό αέριο. Αυτό είναι το ερώτημα. Μιλώντας για μη συμβατικούς πόρους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υποδιαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα ε, πόρων. Μπορούμε να έχουμε ε, άμμο που εμπεριέχει ε, πετρέλαιο, αν θέλετε, που εμπεριέχει το πετρέλαιο. Μπορούμε να έχουμε συστολιθικό αέριο, που το έχουν οι Αμερικανοί. Μπορούμε να έχουμε άλλα είδη αερίου αέριο που προέρχεται φερρυπίν από μη διαπερατά σήματα, ε, διάφορα ειζήματα ε, που εμπεριέχουν μεθάνιο και αυτό είναι σε όλους τους βυθούς των θαλασσών και των ωκεανών ε, και έχουμε και άλλα είδη φυσικού αερίου που εμπεριέχονται σε ανθρακούχα στρώματα. Τώρα θα μιλήσουμε για τα σχιστολιθικά, σχιστολιστικό φυσικό αέριο. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες για να το εξορίξουμε αυτό το αέριο. Τα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αυτού του αερίου μας δείχνουν ότι το σχιστολιθικό αέριο ε, είναι σε μεγάλες ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε άλλες χώρες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική πηγή. Πώς μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών πηγών και πόρων. Ε, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων και των συνεπειών ε, από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Το σχιστολιθικό φυσικό αέριο εμφανίζεται σε μη διαπερατά, σε διαπέρατα πετρώματα και και θα πρέπει να μπορούν όμως να ε, ραγίσουν για να μπορούμε να αφαιρέσουμε τα αέρια οι γεωλογικές παράμετροι θα πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων. Ε, το συνολικό περιεχόμενο σε ανθρακούχο περιεχόμενο και η, μορφή του ορυκτού. Και, και χρησιμοποιούν διαφορετικέ μεθόδους εντοπισμού και εξόριξης, διότι εδώ περνάμε από διαφορετικά στρώματα από ότι όταν ψάχνουμε συμβατικέ πηγέ και χρησιμοποιούμε και διαφορετική τεχνολογία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υδρορογμάτωση χωρί να γνωρίζουμε και ποια είναι η γεωλογική δομή τη περιοχή. Ποια είναι η στρωμάτωση από τα μεγάλα βάθη προς, την επιφάνεια. Η, θα πρέπει να συνδυάζονται διάφορες μέθοδοι, θα πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, κράμα μεταξύ εκμετάλλευσης επιφανειακής, όπου αυτό μπορεί να γίνει, είτε τι δυνατότητα υπάρχει να εκμεταλλευτούμε τα διάφορα φρεάτια και θα πρέπει να κάνουμε ε, ανάλυση και των κομματιών που βγαίνουν από τα φρεάτια. Λοιπόν, να αναφερθούμε τώρα στις, ε, στα διάφορα εδάφη, τα περιέχουν πετρεολεούχα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται ε, τα μόδι πετρώματα αυτά στον Καναδά. Είναι μεγάλες οι και έχει, υπάρχει μεγάλη αύξηση εκμετάλλευση τη αμμόδου πίσας. Έχουν γίνει έρευνες στη Ρωσία, στη Μαδαγασκάρη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και τα αποθέματα, τα διαθέσιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα κέρδη από την εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων ε, είναι πάρα πολύ μεγάλα και η τεχνολογία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική διότι η εκμετάλλευση σε ανοιχτά φρεάτια συνεπάγεται ε, κάποια επένδυση, ε, σημαντικές επενδύσεις. Λοιπόν, αυτή η αμμώδης πίσα περνάει από διάφορες διαδικασίες, ούτω ώστε τελικά να πάρουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αλλά σήμερα αστιαζόμεθα επί, τον, επί του σχιστολίθου, τον πηγών από το σχιστόλιθο, έρευνα και εκμετάλλευση. Τα αποθέματα αυτά υπάρχουν περίπου σε 40 γεωλογικές λεκάνες όλο τον κόσμο, σε αρκετές χώρες δηλαδή και αυτά τα αποθέματα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να εξαχθεί το φυσικό αέριο από το σχιστόλιθο ή το μη συμβατικό αέριο αν θέλετε. Αυτό το σχιστολιθικό αέριο βρίσκεται με διαφορετική τεχνολογία, τα αποθέματα που υπάρχουν σημαντικά και το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα αποθέματα ε, είναι πολύ μεγάλο, είναι ανάμεσα στα 3 και 3,5 χιλιόμετρα βάθος πρέπει να πληρούνται αυτές οι συνθήκες ώστε να μπορούμε να πάρουμε το αέριο. Η παραγωγή στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το ποσοστό μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών πόρων έχει αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ. Με κίτρινο βλέπετε τα μη συμβατικά αποθέματα και με γαλάζιο, με μπλε βλέπετε τα συμβατικά αποθέματα. Η τάση είναι να αντικαθίσταται μια κατηγορία πόρων από την άλλη τώρα μιλώντας για την Ευρώπη, αυτά τα μορφώματα προέρχονται από διάφορες γεωλογικές περιόδους, από 550 εκατομμύρια έτη χρονολογούνται. Υπάρχουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις κάτω χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Νορβηγία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και σε πολλές άλλες χώρες. Σε αυτές τις χώρες γίνεται διερεύνηση για την ύπαρξη των αποθεμάτων και απεδείχθη ότι υπάρχουν τέτοια αποθέματα φυσικού αερίου στα, στους σχηματισμούς που βλέπετε στο κίτρινο, με κίτρινο χρώμα. Αυτά τα μορφώματα έχουν διάφορες ονομασίες αυτά τα, στις διάφορες χώρες, αλλά είναι παρόμοια ε, όσον αφορά τις ιδιότητες που έχουν. Όμως, καμιά φορά δημιουργείται κάποια σύγχυση διότι στην ειδική ορολογία είναι διαφορετική η κατονομασία τους, όμως μιλάμε για αέριο που έχει θερμικές ιδιότητες. Αυτά τα είδη των πόρων πρέπει να πληρούν διάφορες προϋποθέσεις για να είναι δυνατή η εκμετάλλευσή τους. ιδιότητες είναι το μέγεθος των σωματιδίων, ορυκτολογία, οργανικές ουσίες, ένταση, συγκέντρωση, ε, τόπο συγκέντρωσης ε, των οργανικών ουσιών. Ε, αυτό είναι το επίπεδο που διαμορφώνεται το θερμικό αέριο στα 3 χιλιόμετρα περίπου σε σχέση με το βίο αέριο που είναι περισσότερο, είναι πιο κοντά στην επιφάνεια. Γιατί χρειαζόμαστε ειδική μέθοδο ούτως ώστε να εξαχθεί το φυσικό αέριο από αυτά τα μορφώματα, αυτά τα σχήματα τα γεωλογικά. Διότι αντίθετα με το φυσικό αέριο, το παραδοσιακό, το συμβατικό, βρίσκεται στην, ε, στο, στα κενά μεταξύ των σωματιδίων μέσα στα μορφώματα αυτά, σε επίπεδο κρυστάλλων ή σε μικρορογμές. Μιλάμε για μεγέθη της τάξης των μικρών ε, σε πάχος και πρέπει να σπάσουν, να διαραγούν αυτά τα μορφώματα για να αποσπαστεί το φυσικό αέριο. Μετά, σε Έχουμε και το αέριο που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Δεν μπορούσε να ανακτηθεί μέχρι τώρα γιατί ήταν πολύ πιεσμένο. Α, τα μορφώματα από τα οποία αποσπούσαμε του υδρογονάνθρακε είτε σε μορφή πετρελαίου είτε σε μορφή φυσικού αερίου έχουν ποσοστό 30 με 50% ανάκτηση. Οι υπόλοιποι μένουν στα κατάλοιπα. Λοιπόν, μπορεί να ανακτηθεί το αέριο που απομένει αν χρησιμοποιηθεί ε, η σωστή ε, τεχνολογία και έχουμε δευτεροβάθμια ανάκτηση του εναπομένοντος φυσικού αερίου. Οπότε δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτά τα αποθέματα που μπορούν να δώσουν, να συμβάλλουν στην, ε, στις παγκόσμιες, στα παγκόσμια αποθέματα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί που είχαμε και φυσικούς παραδοσιακούς πόρους, συμβατικούς πόρους. Όπως και με το σχιστόλιθο, το συμπαγές φυσικό αέριο ε, μπορεί να βρεθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος Και αυτό λόγω των υδροστατικών συνθήκων ε, που ισχύουν στο υπέδαφος. Μία ιδέα για την εξόριξη αυτών των ουσιών είναι να εγχύεται διοξίδιο του άνθρακος το οποίο μπορεί να λύσει και τα προβλήματα του αερίου του θερμοκηπίου. Διότι το διοξείδιο του άνθρακο, αν συνδυαστεί με νερό, μπορεί να υγροποιήσει αυτέ τι ουσίε και μπορούν να αποσπαστούν και να ανακτηθούν πιο εύκολα. Επειδή κατάγονται τη Ρουμανία και η Ρουμανία είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσα να αναφέρω και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα είδη του φυσικού αερίου και εδώ βλέπετε τις γεωλογικές περιόδους, γεωλογικές περιόδους στις οποίες βρίσκονται αυτά τα φυσικά αέρια και εδώ είναι οι τοποθεσίες στην περιοχή της Ρουμανίας, στα Καρπάθια, σε διάφορους τομείς, στον Μποντλάντ, στο, στην κοιλάδα της Πενωνίας και σε άλλες, ε, σε άλλες λεκάνες και στην, ε, στον εύξηνο πόντο στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχουν γίνει σημαντικές ανακαλύψεις για παραδοσιακό φυσικό αέριο ε, πρόσφατα, για συμβατικό φυσικό αέριο. Άρα έχουμε πολλές δυνατότητες και πληρούνται εδώ πολλές από τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε αυτά τα μορφώματα τελικά να μπορούσαν να παράγουν φυσικό αέριο για καύση. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από τα Καρπάθια, τέτοια πετρώματα από τα Καρπάθια, που πήραμε δείγματα και κάναμε ανάλυση βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Και αυτές οι αναλύσεις δείχνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση των πηγών ε, κάναμε και γεωλογικές δοκιμές για να βρούμε ακριβώς που βρίσκονται αυτές τις ουσίες. Χρειάζεται επιτόπια έρευνα ε, και στις γεωτρήσεις, μέσω γεωτρήσεων κάναμε αυτές τις έρευνες και τελείωσε και ερευνητική φάση. Η φάση των γεωτρήσεων πέρασε, της διερεύνησης, η χαρτογράφηση έγινε ε, και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην εκμετάλλευση, στη φάση της εκμετάλλευσης, διερεύνησης, της πρακτικής διερεύνησης, εξερεύνησης μάλλον και μπορούμε να διατηρηθούμε κατά πόσο αξίζει τον κόπο ε, η όλη προσπάθεια και κατά πόσο το κόστος ε, δείχνει ότι αξίζει η προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια την, ε, περί, την περίοδο της έρευνας, της αξιολόγησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης. Βλέπετε στο γράφημα τι γίνεται με τις χώρες στην περιοχή των Καρπαθίων που δεν έχουν επενδύσει επαρκώς ότι υπάρχουν επίσης και άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ελβετία, οι οποίες χώρες έχουν εντοπίσει ε, αποθέματα. Πρέπει τα πετρώματα αυτά να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και τα αποθέματα χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε ε, περίπου πόσα, τι ποσότητες υπάρχουν και στη ΣΥΠΑ και στη, στην Κίνα προχώρησαν στην φάση της εκμετάλλευσης, έχουν προχωρήσει πιο πολύ. Χρειαζόμαστε λοιπόν να δώσουμε προσοχή στις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών συνεπειών που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η εκμετάλλευση μέσω εξόριξης και η εκμετάλλευση του πετρελαίου δημιουργούν κινδύνους μόλυνσης του περιβάλλοντος και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν μελέτες ε, συνεπιών για το περιβάλλον. Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει τέτοιες αξιολογήσεις. Δεν πρέπει να περιμένουμε για τα πρώτα αποτελέσματα της εξερεύνησης για να αξιολογήσουμε τους κινδύνους. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά που έλεγε ο κ. Όλτμαν δηλαδή ε, στην υδρορογμάτωση που είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση αυτών των πετρωμάτων. Η υδρορογμάτωση είναι κλασική μέθοδος, χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70 αλλά μέχρι τώρα ε, δεν δόθηκε ιδέως προσοχή στις συνέπειες που έχει η υδρορογμάτωση στα ύδατα και όσον αφορά τους σεισμούς, αν έχει και σεισμικές συνέπειες τα ύδατα έχουν κάποια θέση ε, όσον αφορά τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Ε, εδώ βλέπουμε αυτά τα ύδατα τα, στο υπέδαφος που έχουν συγκεντρωθεί με στα πετρώματα που είναι πάνω από το φυσικό αέριο. Τα ύδατα εδώ. Όταν μιλάμε για το νερό που χρησιμοποιείται στην υδρορογμάτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ποσότητες ύδατος απαιτούνται και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα διότι οι αναγκαίες ποσότητες ύδατος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χρησιμοποιούμε ένα μείγμα υδάτων και άμμου 99,5% και 0,5% ε, είναι διάφορες προσθετικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε μια συνταγή αν θέλετε που έχει κάθε εταιρεία ανάλογα με τη γεωλογική δομή των πετρωμάτων και, και στο σημείο που γίνεται η γεώτρηση. Διότι η γεωλογική δομή μπορεί να περιέχει άλατα, άλλες ουσίες, ε, τα πετρώματα τα οποία μπορούν να διαλυθούν φυσικά και αυτό αλλάζει και την, ε, ε, τη σύσταση του νερού που επιστρέφει στην επιφάνεια. Κάποιες από τις ουσίες ε, χρησιμοποιούνται σε καλλιντικά επίσης Έχουμε βαρέα μέταλλα που είναι παρόντα σε επιφανειακά πετρώματα και περιέχονται στα ορυκτά που αποτελούν αυτά τα πετρώματα. Όταν βρέχει πάρα πολύ, σε πιο υγρές περιοχές μπορεί να, να ανέβουν στην επιφάνεια και να βγουν στα πηγάδια των ε, σπιτιών και στα επιφανειακά ύδατα. Ε, και σε αργυλώδη εδάφη μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να περιέχονται βαρέα μέταλλα ε, και σε άλλα πετρώματα τα οποία αποτελούν και την, τον φλοιό ε, της γης, την επιφάνεια. Α, αυτά, αυτές οι συγκεντρώσεις, αυτά τα πετρώματα είναι συνήθως υψηλοί αλλά δεν φτάνουν στα όρια συναγερμού στα οποία πρέπει αν ξεπεραστούν αυτά τα όρια πρέπει να δοθεί προσοχή. Το σύστημα λοιπόν βλέπετε εδώ το υδάτινο που είναι εντελώς κλειστό εκεί που κυκλοφορεί το νερό είναι κλειστό αναφέρθηκε προβληματισμός για ραδιενέργεια κατά πόσο στον άργυλο έχουμε μεγαλύτερη ραδιενέργεια. Κανονικά στο χώμα το αργυλώδες υπάρχει μεγαλύτερη ραδιενέργεια από ό,τι σε άλλα πετρώματα. Και βλέπουμε με το, στο σήμα εδώ, βλέπαμε ακριβώς ε, τι γίνεται με τα πετρώματα. Η υδρορογμάτωση ε, λαμβάνει η χώρα σταδιακά, έχουμε διάφορες φάσεις, ε, μπορεί να δημιουργήσει σεισμικές συνέπειες ε, σεισμούς της τάξης 1 με 2 της κλίμακας Ρίχτερ, έτσι αναφέρεται. Αλλά ε, δεν υπάρχει αντίκτυπος όσον αφορά τα ίδια τα πετρώματα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, αναλύσεις ε, συναρτήσει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, διότι και οι φυσικές σεισμικές κινήσεις του εδάφους διαφέρουν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, κάμπων ε, και σε σχέση με άλλες ε, περιοχές που υπάρχουν άλλου είδους πετρώματα. Ε, Κατακλείδη, υπάρχουν δυνατότητες στην Ευρώπη, θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν όμως θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει σε βάθος μεγαλύτερο από τα 3,5 χιλιόμετρα. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για να εξετάσουμε τι δυνατότητε υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν τελικά μακρηγόρησα και ξεπέρασα τα χρονικά όρια που μου διατίθεντο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που σας υπενθύμησα το χρονικό περιθώριο, αλλά πρέπει να σεβόμαστε, ξέρετε, το χρόνο. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίσκα ζήτησε το λόγο. Α, μικροφώνου. Α, συγγνώμη, έτσι μου είπαν, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εντάξει, δεν πειράζει. Έχω ένα πρόβλημα με αυτές τις δύο εκθέσεις, διότι φαίνεται να διαφέρουν η από την άλλη κάπως προς το περιεχόμενο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι κάτι καινούριο για μας, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το καθεξής, αλλά στην έκθεση του κυρίου Αλπμαν φαίνεται να ε, παρουσιάζονται όλες οι αρνητικές πτυχές ε, του αερίου από σχιστόλιθο. Όποιες ε, αρνητικές πτυχές θα μπορούσε κανείς να βρει. Έχουμε συζητήσει επίσης αυτή τη νέα έρευνα, αυτή τη νέα έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές μας εδώ στο Κοινοβούλιο και φαίνεται ότι η επικαιροποιημένη δική σας εκδοχή δεν αλλάζει και πολύ τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη το διοξίδιο του άνθρακα το οποίο εκλείεται κατά την παραγωγή αερίου χιστόλιφο. Υπάρχουν κάποια ευρήματα αντιφατικά αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι το φυσικό αέριο το οποίο έρχεται μέσω Ρωσίας εκλείει, εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με την παραγωγή αερίου χιστόλιφο. σας κατάλαβα καλά. Αυτά νομίζω λένε και τα τελευταία στοιχεία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάλι λένε κάτι διαφορετικό, ότι το αέριο όπως χιστόλιθο δεν παράγει. Η εξόριξη αερίου δεν παράγει σημαντικές ποσότητες οξυδίου του άνθρακα. Θα ήθελα λοιπόν και από τους δυο σας να κάνετε μια αντιπαραβολή των στοιχείων σας και να δούμε τι συσχετισμοί υπάρχουν. Κύριο Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, ε, έχουμε κάποιο χρόνο για συζήτηση. Με απογοήτευσε λίγο η παρουσίαση. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε λάβει υπόψη των πορισμάτων και δεν έχουν αλλάξει έκτοτε. Η εκτίμηση επιπτώσεων που προτείνει η ιδιωτική εταιρεία του κ. Άλτφαν δεν επιβεβαιώνεται από κανένα, καμία άλλη μελέτη που γνωρίζω να έχει γίνει είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι κυβερνήσει, από τον κλάδο, από τη βιομηχανία, από ακαδημαϊκού. Περίεργο αυτό. Για πρώτη φορά σε μια μελέτη βλέπουμε ε, να αξιολογείται ω υψηλό ο κίνδυνο. Ε, είναι η μόνη τέτοια μελέτη που ξέρω να έχει τουλάχιστον αυτή την κατάληξη, αυτά τα πορίσματα. Και είναι κρίμα πραγματικά που δεν λαμβάνει υπόψη καμία από τι θετικέ εξελίξει, ιδίω ό,τι αφορά τη χημική διαφάνεια ε, στη βιομηχανία. Πρόκειται για μια τεράστια εξέλιξη στην έκθεση που ψηφίσαμε στην Επιτροπή ΕΝΒ και στην Επιτροπή ΙΤΡΕ. Τα λέμε όλα αυτά και ελπίζουμε να είναι και ε, μια καλή είδηση και για τη βιομηχανία και για τους πολίτες. Αλλά στην έκθεση αυτή δεν τα περιλαμβάνεται. Και ακόμη κάτι που με εξέπληξε, ακόμη περισσότερο μάλιστα, εδώ και 1,5 χρόνο μελετούμε τις νέες πληροφορίες ε, για την ε, εξόριξη φυσικού αερίου πασχιστόλτα. Στην Πολωνία, στην Πομερανία συγκεκριμένα, σε ένα Ινστιτούτο, έγινε η πρώτη και μόνη μέχρι στιγμή συνεκτική μελέτη επιτόπου, όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος ε, της υδρορογμάτωσης και γίνονται πάρα πολλά, δίνονται πολλά στοιχεία για το αποτύπωμα άνθρακα και την έκκληση σε εκπομπές, όλα αυτά. Είναι πολύ πλοκή η τεχνολογία. Σίγουρα πρέπει να δούμε αν πληρούνται τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμω αυτή η μελέτη την οποία σα ανέφερα δεν αναφέρει ούτε μία φορά στην λεγόμενη επικαιροποιημένη σα αυτή μελέτη. Η πρόεδρο, έχετε δύο λεπτά να απαντήσετε. Κύριε Αναστασιώστη, αφορά το ερώτημά σας. Έχω ε, να σας δώσω τις εξής απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ε, να έχει κανείς γνώση του πώς συλλέγονται τα στοιχεία. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, εάν τα αποθέματα μεθανίου αυξάνονται στην Ευρώπη, τότε είναι σαφές ότι θα μειωθούν οι εισαγωγές. Ίσως αυτό να μην είναι και τόσο καλό και αυτούς που αυτή τη στιγμή εξάγουν σε πολύ ψηλέ τιμές μεγάλες ποσότητες αέριου. Θα πρότεινα λοιπόν να γίνει μια συγκριτική μελέτη, μια συγκριτική ανάλυση για να δούμε τι δυνατότητες προσφέρουν οι συμβατικοί και μη συμβατικοί πόροι και αν τα αποτελέσματα της εξόριξης με την τεχνική της υδρορογμάτωσης που μιλάμε για τη δεκαετία του 70 ε, δεν θα πρέπει να αναλυθούν, να αναλυθούν δύο-τρεις περιπτώσεις τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι εκατοντάδες ε, γεωτρήσεων λαμβάνουν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ε, είπα συγγνώμη, και υπήρξαν και ατυχήματα. Θα πρέπει τα πράγματα να τα εξηγούμε με διεξοδικό και πλήρη τρόπο. Θα πρέπει να αναλύσουμε και ε, τι προκύπτει σε ό,τι αφορά τη ρήπανση των υδάτων και θα πρέπει να αναλύσουμε και τον κίνδυνο σεισμικών κινήσεων. Αυτό το επιχείρημα όταν το ακούνε οι γεωλόγοι γελάνε. Πρέπει να γίνουν κάποιε αναλύσει, γιατί μόνο έτσι θα έρθουμε πιο κοντά στη λύση του προβλήματο. Αναφέρατε επίση το ζήτημα τη παρακολούθηση, του ελέγχου. Εάν ε, πονήσουμε ένα νόμο που θα απαιτεί να υπάρχει επιτόπου παρακολούθηση και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, τότε πάλι νομίζω ότι θα πλησιάσουμε την αλήθεια. Ευχαριστώ και ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Δηλαδή εμένα είναι να αναλύσω από επιστημονική πλευρά ε, του κινδύνου. και σε ποιο βαθμό μπορούμε να συγκρατήσουμε, να ελέγξουμε αυτού του κινδύνου. Ό,τι αφορά τώρα την ισορροπία του ισοζύγιο δεξιδίου του άνθρακα, έχετε δίκιο ότι η μελέτη που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία δημοσιεύθηκε πριν από τρει εβδομάδε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ισορροπία ε, είναι καλύτερη σε σχέση με την περίπτωση εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Εγώ προσπάθησα να τονίσω το εξή. Υπάρχει μία προειδοποίηση, κάτι πρέπει να προσέξουμε εδώ. Τα παρουσίασα τα αποτελέσματα, υπάρχει όμως ένας περιορισμός, ένα caveat. Ουσιαστικά είδαμε μηδέν ουσιαστικά μηδενικό περιεχόμενο ε, στο αέριο ε, που εξάγεται σε διεξίδιο του άνθρακα. Η Exxon Mobile τώρα, στις πληροφορίες που μας έδωσε σε σχέση με τις λίγες υδρορογματώσεις που έχει διεξαγάγει λέει ότι η περιεκτικότητα ε, στο αέριο το οποίο εξάγεται, σε, η περιεκτικότητα σε διοξιδάκι είναι της τάξης 3,5 3 ε, ε, έως 5 και εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται. Έχουμε επίσης στο Μίσιγκαν ένα πεδίο γεωτρήσεων, πολύ παλιό, και εκεί η περιεκτικότητα περιβαίνει το 30%. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς εδώ, αναλύουμε το χειρότερο σενάριο, δηλαδή υποθέτουμε ότι θα είναι 30% υπερεκτικότητα του διοξιδίου του άνθρακα στο αεροπεξοέστη για να δούμε τι επιπτώσεις έχει αυτό. Θέλω να σας ε, επαναλάβω το εξή. Πρώτα απ' όλα έχουμε ε, την τεχνολογία, έχουμε τη διαχείριση για να μειώσουμε τις εκπομπές το θέμα είναι αν μπορούμε να επηρεάσουμε την περιεκτικότητα του αερίου που ε, εξορίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στην παρουσίαση των αναφορών. Πρώτη αναφορά συγκεκριμένα ελήφθη από την Γαλλία και την ε, κατέθεσε η κυρία Ντανιέλ Φαβάρη. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση από την κυρία Φαβάρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Στην πάλη ε, που διαξάγουμε καθημερινά προσπαθούμε να δράσουμε για το περιβάλλον, τον πλανήτη και την απειλούμενη βιοπικιλότητα. Κανείς δεν αγνοεί ότι η θέρμανση είναι κατά 90% ανθρώπινης προέλευσης και αυτό θα δημιουργήσει τεράστιες ε, ε, αλλαγές στη βιόσφαιρα και την ανθρωπότητα. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους ηγεμόνες μας, τους ηγέτες μας μάλλον ότι οι ανάγκε του παρόντο δεν πρέπει να θέσουν εν κινδύνο την δυνατότητα του μέλλοντος να ικανοποιήσει τις δικέ του ανάγκες. Η μάχη αυτή γίνεται για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της ε, εκμετάλλευσης που ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει ασφαλή με οποιοδήποτε τεχνική των αερίων και των, ε, του πετρελαίου από το σχιστόλιθο. Αν η γαλλική κυβέρνηση εμείνει στην απαγόρευση της ε, υδρορογμάτωσης. Θέλω να κάνω μια παρένθεση γιατί πολλοί μιλάνε για υδρορογμάτωση. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για νέες μορφές ε, υδρορογμάτωσης με το διοξείδιο του άνθρακος ή με ήλιο όπως είπε κάποιος προηγούμενος. Αλλά δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ για αυτήν την εξόριξη βιομηχανική διαδικασία που είναι οικολογικά αποδεκτή οικονομική κατάσταση δεν θα επιληθεί με αυτήν την ε, ενέργεια που είναι παρακόλληση στην ουσία. Δεν είναι ε, βιώσιμη αυτή η ενέργεια διότι η δημιουργία θέσεων εργασίας με, τις, ε, με τα με τα ορυκτά καύσιμα είναι μύθος. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε όλες τις ε, εναλλακτικές που παρουσιάζονται. Μας είπαν ότι θα αξιοποιήσουμε μόνο το 20% του αερίου και του πετρελαίου από το σχιστόλιθο και ότι θα μειωθεί σύντομα η παραγωγή. Η υδρορογμάτωση είναι τεχνητή και αυτή η διαδικασία προκαλεί μία ανεπίστρεπτη διαδικασία εισαγωγής ε, αερίου που θα κρατήσει ανά δεκαετίες, κατά δεκαετίες, για δεκαετίες. Και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα έχουμε τεχνική που θα μας επιτρέψει να επανέλθει ο σχιστόλτος στην αρχική του κατάσταση. Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες, ιδιαίτερα διότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνο και έκκληση διοξιδίου του άνθρακο. Μία άλλη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Μπάουντερ από 27 επιστήμονε αποδεικνύει ότι οι εκκλήσει και οι μεθανίου έχουν ένα ε, δυναμικό θέρμανση του πλανήτη 25 φορές περισσότερο από το δεξί του άνθρακος. Όπως ξέρετε πολύ καλά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και με τους ε, σωλήνες και καταλαβαίνετε ότι τα αέρια αυτά είναι ιδιαίτερα πτυτικά και μπορεί να συνεχίσουν να βγαίνουν και μετά το κλείσιμο των φρεατίων. Οι 25 σεισμογράφοι που παρακολουθήθηκαν στο Τέξας για δύο δεκαετίες μας επέτρεψαν να διαπιστώσουμε χαμηλού επίπεδου σεισμού, αλλά το επίκεντρό του είναι ακριβώ στι περιοχέ όπου είχαν γίνει μεγάλε υδρορογματώσει. Γιατί όποια και να είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται, η υδρορογμάτωση αποσταθροποιεί το υπέδαφο. Όπω είπε η Κομισιόν, δεν υπάρχει καμία νέα προδιαγραφή που να είναι αναγκαία για να ρυθμίσουμε αυτή την εκμετάλλευση. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής ρυθμιστική νομοθεσία είναι δύσκολη γιατί βασίζεται κυρίως στα προϊόντα και εδώ αναφέρομαι και στην προηγούμενη εκδοχή της έκθεσης γιατί ήδη έχουν σημειωθεί εννέα μεγάλα κενά στην αποτίμηση που κάνουμε και δεν αναφέρονται στις οδηγίες που αφορούν τον περιορισμό των εκπομπών από διάφορους ρηπαντές στην ατμόσφαιρα η δραστηριότητα από την εκμετάλλευση του αερίου και του πετρελαίου από το σχιστόλιθο. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε ιδιαίτερα το περιβάλλον μας, να συμφωνήσουμε με τις προτροπές του ΟΣΑ, πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε το περιβάλλον, ότι η μόλυνση είναι πολύ πιο ακριβή από το σεβασμό του περιβάλλοντος, να λάβουμε υπόψη τις συμβουλές του Γαλλικού Συμβουλίου ε, για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, το στόχος μας πρέπει να είναι να υπάρχει μηδέν επίπτωση. Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυτών που παράγουν και αυτών που ρυθμίζουν. Δεν πρέπει λοιπόν επίσης να υπάρχουν ε, επιδοτήσεις ε, για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει να υποχρεώσουμε τους, τις εταιρείες που εργάζονται σε αυτό το τομέα να μας χορηγήσουν επαρκείς εγγυήσει και οικονομικές αλλά και επί της ουσίας για να καλυφθεί οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από την δραστηριότητά τους και να υπάρχει νομική ασφάλεια στους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές. Διότι εφόσον υπάρχει άμεση απειλή για περιβαλλοντική ζημία, κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει μια αρμόδια αρχή που είναι υποχρεώσει τους εκμεταλλευόμενους να πάρουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα ούτω ώστε να μπορέσουμε μετά να καλυφθούν τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από την δραστηριότητα αυτή. Είναι λοιπόν βασικό το θέμα των ε, ασφαλιών. Όπως βλέπουμε υπάρχουν νομικές αβεβαιότητες, αν και η έννοια της οικολογικής ζημίας ήδη υπάρχει ομολογία μέσω της δίκης του Έρικα, πρέπει να καθορίσουμε σε τι επίπεδο πρέπει να υπάρξει απομόλυνση για να επανέλθουν οι περιοχέ στην ε, κατάσταση που ήταν πριν, ιδίω αν έχουν υπάρξει διαδοχικές ε, βιομηχανικές Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, που δεχτήκατε την αναφορά μας. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή Ένδη που καλεί σε σόφρονα αντιμετώπιση και καλεί να υπάρξει ε, λεπτομερής ανάλυση στον τομέα αυτό ούτω ώστε να παλέψουμε κατά της ε, χειροτέρευσης των εδαφών μας. Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Χρήση του Άνθρακα και στις 19 Φεβρουαρίου θα το ξανασυζητήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο για ε, βιώσιμη οικολογική ανάπτυξη διότι δεν είναι απλώς ε, το μέγιστο του πετρελαίου, αλλά τα δικά μας όρια που έχουμε φτάσει. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχουν δύο άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα από τη Ρουμανία. Πρώτη είναι από την οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώματα. Η οργάνωση αυτή είναι κατά της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης του ε, σχιστολιτικού αερίου στη Ρουμανία, διότι μπορεί να καταστρέψει τους υδροφόρους ορίζοντας τις παράκτες αυτές τις ρουμανικές περιοχές και ζητούν την ε, αναστολή του ε, προγράμματος ε, αυτού μέχρι να υπάρξει δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Η δεύτερη αναφορά είναι του κ. Βασίλε Στάν που έχει αντίρρηση στην εκμετάλλευση του σχιστολιτικού αερίου τονίζοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι υδρογονάνθρακες που προκύπτουν από αυτά τα πετρώματα δημιουργούνται κατά εκατομμύρια χρόνια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ανισχύει λοιπόν για τους κινδύνους που προκύπτουν από την εξόριξη αυτών των αποθεμάτων και αναφέρει ενδοκρινολόγους ε, του ε, Ιατρικού Ινστιτούτου Κορνέλ ε, στις Ηνωμένες, στις Νέα Υόρκη, που καλούν να υπάρξει ένα μορατόριο μέχρι να εξεταστούν οι επιπτώσεις. Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας. Πρέπει να υπάρξει moratorium στην διερεύνηση και εξόριξη σχιστολιτικού αερίου. Για αυτές τις αναφορές έχουμε την ε, νομική ανάλυση ε, της κυρίας Μάρθας Μπαγεστέρος. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μάρθα Μπαγιστέρος. εκπροσωπώ το Μιλιέ, μια εταιρεία που αποτελείται από δικηγόρους και ανθρώπους που την πολιτική έχει έδρα στις και διεξάγουμε αναλύσεις νομικού περιεχομένου, πολιτικού περιεχομένου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας ζήτησε την άποψή μας σε σχέση με ορισμένε νομικές πτυχές ε, των αναφορών. Εξετάσαμε κυρίως τις αναφορές που μας δόθηκαν στα γαλλικά, τις γαλλικές κυρίως δηλαδή, και αυτό που κυρίως μας απασχολήσει είναι το ενδεχόμενο ενός νέου κανονισμού μέσου μιας διάταξης δηλαδή καινούρια σε σχέση με το αεροποσχιστόλιθο. Ε, έχουμε τις οδηγίες για, μάλλον τις ε, οδηγίες πλαίσιο για τα ύδατα, περιβαλλοντικής, εκτίμηση περιβαλλοντικών και επιπτώσεων. Και αφού θα μιλήσουμε για ένα νέο μέσο που θα απαγορεύει δραστηριότητε εξόριξη και σχιστολιθικού αερίου, θα κάνουμε κάποια συμπεράσματα. Όπω βλέπετε, υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Στι αναφορέ, μία από τι πτυχέ που τίθεται είναι ότι δεν υπάρχει πλήρης και αναλυτική μελέτη και εξέταση του νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το πλαίσιο η δυνατότητα, η ανάγκη ειδική ε, διάταξης ή νομοθετήματος για το σχιστολιθικό αέριο είναι απαραίτητη. Οι αναφέροντες ως προς το σημείο αυτό τόνισαν την νομοθεσία για τις εξορρεκτικές δραστηριότητες για τα ορυχεία και ε, πρότεινα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει νέα νομοθεσία βασιζόμενη σε αυτήν για τα ορυχεία και επίσης υπάρχουν ε, και κάποιες ε, προτάσεις σε ό,τι αφορά την άντληση νερού, όπως αυτή προβλέπεται στην νομοθεσία, επιπτώσεις στο νερό, λόγω του κινδύνου που προκύπτει από τη χρήση χημικών ουσιών, οι αναφέροντες μεταξύ άλλων ανέφεραν την ανησυχία τους γιατί δεν μπορεί η οδηγία για την εξολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αντιμετωπίσει κάποιες πτυχές που άπτονται της εξόρυξης αερίου από σχιστόλιθο. Δεν υπάρχει επίσης συνέπεια, συνεκτικότητα μεταξύ της ε, ερευνητικής γεώτρησης και της εκμετάλλευσης αερίου από σχιστόλιθο. Κάποια ζητήματα επίσης που της ενεργειακής πολιτικής, ε, της ε, του περιορισμού της Χρυσάθακα, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα λάβαμε υπόψη και τα βλέπετε στις διαφάνειες. Δεν υπάρχει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθεσία η οποία θα ασχολείται ειδικά με το αεροποσχιστόλι. Αυτό είναι σαφέ και βέβαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί στην παρούσα φάση το κατά πόσο το τρέχον ε, νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ορθό, είναι αυτό το οποίο θα καλύψει ε, με τον κατάλληλο τρόπο όλες τις δραστηριότητες που άπτονται του σχεστολικού ΕΡΤ. Τρεις δημοσιεύσεις έχουμε, τις ανέφεραν οι προλαλήσαντες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κάποιες τεχνικές οικονομικές πτυχές και υπήρξαν και δύο διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν που θα οδηγήσουν στη δημοσίευση δύο ακόμη εκθέσεων που θα εξετάζουν την εθνική νομοθεσία και θα προβαίνουν σε περαιτέρω εκτιμήσει ε, τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συγκεκριμένα θα εξετάζουν το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα πλαίσιο ε, διαχείρισης κινδύνου για το αεροποσχιστόλιθο. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή αυτές τις εκτιμήσεις ε, διανεργεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ορυχεία. Δεν υπάρχει ένα πλήρες πλαίσιο Φυσικά υπάρχουν τέσσερις οδηγίες που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές δραστηριότητες, δύο εκ των οποίων αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Δεν είναι δηλαδή ε, διατάξεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην προκειμένη περίπτωση. Δύο όμως θα μπορούσαν να είναι αυτή που αφορά τα ε, απόβλητα και απορρίμματα το 2006. Εγκρίθηκε και η δεύτερη αφορά τις αδειοδοτήσεις ε, για την παραγωγή δρογοναθράκων. Η πρώτη οδηγία, West Mining Directive, για, την, ε, για τα απόρριτα, ε, απαιτεί την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία δίνει για την ανέγερση, τη διατήρηση, τη διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων. Απαιτεί επίσης από αυτές τις μονάδες να έχουν σχέδιο διαχείρισης να έχουμε συστήματα ασφαλείας, αλλά και την, την, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ε, την κατάρτιση εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων διαχείρισης. Αν χρειαστεί επίσης, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαθέσιμες τεχνικές. Αυτά τα συστήματα, ή μάλλον αυτή η νομοθεσία, καλύπτει μόνο τη διαχείριση των αποβλήτων από ε, εξορρυκτική δραστηριότητα, όχι την εξόριξη και την εκμετάλλευση αέριο όπως στόλιθο. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι πλήρης η νομοθεσία αυτή. Τώρα, η οδηγία του 94 για την ε, διοδότηση ε, παραγωγής ε, δρόμων θράκων. Εκεί θεσπίζονται κάποιοι κανόνες για τις συγκεκριμένε εγκρίσεις διοδοτήσεις, όπου τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κάποιους όρους στις, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αυτών των αδειών με κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό όμω είναι μόνο επιλογή για τα κράτη-μέλη. Δεν υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να το πράξουν. Είναι προαιρετικό. Επομένω, δεν είναι βέβαιο ότι θα το πράξουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτές οι δύο οδηγίε δεν είναι πλήρεις, είναι λυπεί και δεν μπορούν να παράσχουν το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για τα ορυχεία και για την παραγωγή δραπαναθράκων. Μία επιλογή που θα είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εγκρίνει ένα νομοθέτημα το οποίο θα καλύπτει τις υπόλοιπες πτυχές. Το Κοινοβούλιο στις εκθέσεις του και συγκεκριμένα στην έκθεση που θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο, ο επισημένος μέσα από τις πτυχές αυτές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως για παράδειγμα είναι η ταυτοποίηση ε, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Ποιες είναι αυτές ε, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ποιοι τις ε, αναπτύσσουν και τις χρησιμοποιούν, ενώ επίσης περιλαμβάνει και κάποιες απαιτήσει για την κατασκευή του φρεατίου, που δεν καλύπτεται ε, από τις ευστάμενες δύο οδηγίες αυτή η πτυχή. Όπως σας είπα, οι απαιτήσει σχετίζονται με τις μονάδες ε, που εξεργάζονται τα απόβητα. Σε ό,τι αφορά τώρα την επεξεργασία θερμοκηπιακών αερίων από ε, την εξόρυξη αεροποσχεστόλυφα, εκεί υπάρχουν κάποια κενά. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για, τους, ε, για τις επιχειρήσεις να αναφέρουν το πώς ε, αντιμετωπίζουν μετά πώς επεξεργάζονται τα αέρια θερμοκηπίου. Στην ε, οδηγία ITS e περιλαμβάνεται το μεθάνιο, αλλά δεν περιλαμβάνει η δραστηριότητα της εξόρυξης ε, του αερίου από σχιστόλιθο. Οπότε δεν είναι βέβαιο κατά πόσον οι βιομηχανικές εκπομπές καλύπτουν τις δραστηριότητες παραγωγής ε, φυσικού αερίου από σχιστόλιθο. Και να λοιπόν και εδώ. Τώρα να περάσουμε στην ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Η οδηγία αυτή είναι σαφές ότι επιβάλλει υποχρέωση στα κράτη-μέλη να πετύχουν την καλή οικολογική και χημική κατάσταση των υδάτων. Μεταξύ αυτών λοιπόν να αποφύγουν, να, αποτραπεί, να αποφευθεί η επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων Περιλαμβάνονται εδώ και βέβαια οι της εξόρυξης αερίου από σχιστόλιθο. Δεν προβλέπονται όμως τα σχετικά με την υδρορογμάτωση. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της και τεχνική. Υπάρχουν επίσης κάποιες παρεκκλήσεις ε, που θα ήταν δυνατές ε, δυνάμεις οδηγίας πλαίσιο για τα υδατά για τους ελέγχους παραδείγματος που απαιτούνται για την απάντηση ε, νερού. Από αυτές τις εξαιρέσεις παρεκκλήσεις ε, από τους ελέγχους, μάλλον αυτοί, αυτές οι παρεκκλήσεις είναι δυνατές μόνο αν η δραστηριότητα αποδειχθεί ότι δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο. Έχουμε δει λοιπόν το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, τι επιπτώσεις θα είχε η εξόριξη φυσικού αερίου όπως για το περιβάλλον. Αυτό το άρθρο 11 λοιπόν 3ε τη οδηγία για τα ύδατα είναι εφαρμοστέο στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, η οδηγία για τα πήγια ύδατα δεν επικεντρώνεται παραστής αδειοδοτήσει την χρήση των υπογείων άρα δεν είναι εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Υπάρχει και μία ανασφάλεια, νομική ανασφάλεια, σε σχέση με αυτήν την οδηγία πλαίσιο για τα είδη. Στο άρθρο 11.3 συγκεκριμένα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί άδεια για έγχυση νερού, το οποίο περιέχει ουσίες από εξορρεκτική δραστηριότητα, από παραγωγή υδρογονανθράκων. Αυτό το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα σημείο μας στο οποίο κάνει κάποιες διευκρινήσεις για τις ε, άδειες αυτές, ότι δεν είναι οι άδειες δηλαδή που απαιτούνται για την υβρορογμάτωση, ωστόσο δεν είναι βέβαιο από νομικής πλευράς ε, τι συμβαίνει. Μιλάμε για μια ερμηνεία απλά. Δεν έχει δημοσιευθεί ένας νόμος. Ερμηνεύονται κάποιες διατάξεις. Νομίζω ότι αυτά χρήσουν περαιτέρω διευκρίνησης στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας. Οδηγία ΕΠΕ, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτή την οδηγία υπάρχει απέτηση για τη διεξαγωγή τέτοια ε, εκτίμησης εξολογικών επιπτώσεων για τις δραστηριότητε του παραρτήματος 1. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τα κράτη-μέλη για όσε δραστηριότητες δεν είναι καταγεγραμμένε στο παράρτημα 1 να αποφασίσουν και να ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη ορίζοντας τα κριτήρια και τα κατόφλια για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μελέτη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα, στο παράρτημα 1, για την ε, εκμετάλλευση αερίου και υδρογονανθράκων, υπάρχει ένα κατόφλιο οποιοδήποτε έργο, οποιοδήποτε project αποσκοπεί στην εξόρυκτη 500.000 κυβικών μέτρων την ημέρα, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βέβαια, τα έργα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο, όπως το φθάνουν το κατόφλι αυτό σω όντω υπάρξουν αποκλίνούσε ερμηνείε από τα κράτη-μέλη για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα να ότι θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας ώστε η κατάσταση να υπαρξει τροποποιηση τη σχετικη νομοθεσια ωστε η κατασταση να ξεκαθαριστει και στο παράρτημα 1 να περιληφθεί η παραγωγή φυσικού αερίου από στι σχετικέ δραστηριότητε, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι είναι υποχρεωτικό, υπάρχει υποχρέωση για διενέργεια ΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια συμμετοχή και τη διαβούλευση. Έχουμε την σύμβαση του Άρχους από το 2001. Έκτοτε και συγκεκριμένα το 2003 εγκρίθηκε η σχετική οδηγία για να τροποποιήσει την οδηγία ε, για τη μελέτη των επιπτώσεων ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι να μπορεί να υπάρχει δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για έργα τα οποία απαιτούν τη διενέργεια μελέτης αντικτύπου. Έχουμε τρεις πυλώνες σε αυτή τη σύμβαση άρχους. Πρόσβαση στι πληροφορίες, δημόσια συμμετοχή και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και η οδηγία αυτή πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά μόνο στα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη δημόσια συμμετοχή. Επειδή δεν είναι απόλυτα σαφές κατά πόσον ε, τα έργα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την υποχρέωση για την ενέργεια μελέτη σε επιπτώσεων, πρέπει κάποια πράγματα να διευκρινιστούν. Έχουμε και την οδηγία για τα ορυχεία που προβλέπει δημόσια συμμετοχή, αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με την άδεια εκμετάλλευση ή λειτουργία τη ε, μονάδα επεξεργασία των αποβλήτων. Άρα η νομοθεσία που προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού, τη δημόσια συμμετοχή σε έργα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή φυσικού αερίου όπως δεν είναι ξεκάθαρη. Και νομίζουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί αν υιοθετηθούν νέες διατάξεις στο πλαίσιο της φυστάμενης νομοθεσία. Έχει προταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει νομοθεσία που θα απαγορεύει τις δραστηριότητες εξόριξης φυσικού αερίου από σχιστόλιθο. Υπάρχουν τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά, βιομηχανικά ζητήματα. Έχει εγκριθεί νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιβάλλει την εφαρμογή ε, των εφαρμοστέων διατάξεων, αλλά μπορεί και να τις τροποποιήσει τις διατάξεις αυτές. Ωστόσο, με βάση τη συνδίκη της Λισαβόνας, εγκρίνεται πλέον ένα νέο άρθρο για τη ρύθμιση της ενεργειακής πολιτικής. Και ένας από τους στόχους του άρθρου αυτού, συγκεκριμένα το άρθρο 194, είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια της ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια. Επομένως, αυτή η νομοθεσία για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα είχε ως στόχο κατά πάσα πιθανότητα ακριβώς την επίτευξη αυτού του στόχου θα ενέπεται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό το άρθρο όμως απαιτεί όποια μέτρα επηρεάζουν την επιλογή των κρατών μελών για το ενεργειακό μείγμα, πηγές δηλαδή και εφοδιασμό να μην μπορούν να ε, εγκριθούν επειδή άπτονται τη εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Η νομοθεσία που θα απαγόρευε την παραγωγή φυσικού αερίου θα κατέπιπτε ή θα ερμηνευόταν ως βασιζόμενη νομικά σε περιβαλλοντικές διατάξεις, το άρθρο 192 δηλαδή της συνθήκης, οπότε έτσι θα μπορούσε να εγκριθεί, επαναλαμβάνω δυνάμει το άρθρο 192 αν εγκριθεί, ή το 191. Οι αλλά είναι μάλλον απίθανο κάτι τέτοιο, διότι δεν υπάρχει διάταξη νόμος που ε, δεν θα εμπει... Ε, που θα ρυθμίσει τα ενεργειακά και δεν θα εμπίπτει στον ενεργειακό χάρτη. Δεν νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει νομοθεσία για την απαγόρευση του σχιστολιτικού φυσικού αερίου, γιατί αυτό θα επηρεάσει την πρόοδο των κρατών μελών. Ωστόσο, έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει νομοθεσία που θα επιβάλλει όρους με βάση περιβαλλοντικές παραμέτρους σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του αερίου από σχιστόλιθο. Τέτοια μέτρα μπορούν να υιοθετούνται είτε με ομοφωνία, εάν θεωρηθεί ότι πέρασαν σημαντικά τα κρατη την επιλογή του συγκεκριμένα, και αν θεωρηθεί ότι τα μέτρα δεν επηρεάζουν σημαντικά, αλλά μόνο κατά κάποιο βαθμό, σε κάποιο βαθμό την επιλογή των κρατομέλων, μπορεί ε, τα μέτρα αυτά να υιοθετούνται με την απλή διαδικασία της, την κανονική διαδικασία της συναπόφασης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πολιτικής, Α, να φτάσω στα συμπεράσματά μου. Για το τρέχον πλαίσιο πολιτικής λοιπόν, είναι σαφές ότι η τρέχουσα νομοθεσία έχει κενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εκτιμήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ποιο θα ήταν αυτό, υπάρχουν επιλογές, διάφορες πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ή ίσως και μια ε, νέα νομοθεσία για τις εξωτερικέ δραστηριότητες. Υπάρχει ενωσιακή αρμοδιότητα για την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας και την επιβολή περιβαλλοντικών όρων, ίσως όχι όμως αρμοδιότητα για απαγόρευση της δραστηριότητας αυτής. Και επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει η τεχνολογία αυτή πρέπει να εκτιμηθεί με στόχο την εξορρόπηση διαφορετικών στόχων. Αφενός την οικονομική και την ενεργειακή ασφάλεια και αφετέρου περιβαλλοντικοί στόχοι πρέπει να πληρούνται. Στόχοι απανθράκωσης, δηλαδή περιορισμού τη χρήση του άνθρακα ή αύξηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μποστινάρου τώρα. Ευχαριστώ, Ερήτηνη Πρόεδρος. Ε, έχω ένα πρώτο συμπέρασμα. Έχοντας δύο επιστήμονες που παρουσίασαν τις θέσεις τους με αντικρούμενες θέσεις, αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι και πόσο επίκαιρη ήταν η ιδέα της Επιτροπής μας να διοργανώσει αυτή την ακρόαση. Δραματικά απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό. Να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το αναγκαία θεσμικά και νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με το αέριο από το σχιστόλιθο. Θα στραφώ στα ρουμανικά, διότι έχουμε μία αναφορά από τη Ρουμανία και θέλω να μιλήσω και για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στη χώρα μου. Θα μιλήσω ρουμανικά. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, βρήκα ότι ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις. Η μία, ανεφόρον απόρριψη της ιδέας της εκμετάλλευσης στο φυσικό αερίο όπως χιστόλιθο, που αυτή εδράζεται επί επιστημονικών επιχειρημάτων, τα οποία επιχειρήματα δεν είναι πολύ αναλυτικά, και από την άλλη πλευρά, ανεφόρον υποστήριξη για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, που εκφράζει τις απόψεις του πολύ ισχυρού βιομηχανικού λόμπι που αρνείται όμως ε, επιστημονικά στοιχεία και ιατρικά στοιχεία. Η αλήθεια όπως πάντα βρίσκεται κάπου στη μέση. Και η συζήτηση που γίνεται σήμερα το επιβεβαιώνει αυτό. Ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να συναγούμε, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είτε ζουν στη Γαλλία, είτε ζουν στη Ρουμανία, είτε ζουν στη Βουλγαρία, έχουν το δικαίωμα να προβληματίζονται, να ανησυχούν, διότι τους λείπουν οι πληροφορίες. Ε, ανησυχούν διότι ο διάλογος μεταξύ των δημοσίων αρχών και των διαφόρων κοινοτήτων ε, απουσιάζει. Ανησυχούν διότι οι πολυεθνικές εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα και την εξόριξη πολύ συχνά αρνούνται τον διάλογο με την κοινότητα. Πάρα πολύ συχνά οι συμβάσεις ε, για τις αναθέσεις είναι ε, διαβαθμισμένες, όπως συμβαίνει στην Ρουμανία. Πώς μπορούμε λοιπόν αν έχουμε απόρριτες συμβάσεις να έχουμε διαφάνεια. Το πρώτο μου συμπέρασμα είναι ότι εδώ στην Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους πολίτες και τις κοινότητες και τα συμφέροντά τους και θα πρέπει να επιβάλλουμε τη διαφάνεια και για τα κράτη-μέλη και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που ήθελα να σας αναφέρω είναι το εξής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν, παρουσιάζονται ε, στα ειδικά βιβλία. Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε αυτά με έναν τρόπο φθηνό και επιφανειακό που χαλιναγωγείται από τους μεγάλους παραγωγούς φυσικού αερίου που θα διατηρήσουν το μονοπόλιο τους στην αγορά. Είμαι πεισμένο ότι οι πολυεθνικές του φυσικού αερίου δεν είναι αθώες, δεν είναι άγιοι. Αλλά να λέμε ότι τα επιστημονικά κείμενα δείχνουν που δείχνουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι καταστροφές ε, εμπνέονται από αυτά τα επιχειρήματα είναι κάτι απαράδεκτο. Και υπάρχει και κάτι άλλο που μας είπαν οι εκπρόσωποι της εταιρεία συμβούλων. Είναι ότι υπάρχει ανάγκη να θετηθεί πλήρης λεπτομερής ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτό για να καλυφθούν οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών υπάρχουν και προσδοκίε και από τα κράτη-μέλη. Θέλουν να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τι ενεργειακές πηγές. Και το μονοπόλιο του φυσικού αερίου εκεί τίνει να δημιουργήσει κινδύνους λόγω της αυξήσεως του πολύ ακριβού λογαριασμού που δίνει στους πολίτες για την ενέργεια, των πολύ ακριβών τιμών. Ε, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει θεσμικός διάλογος με τις επιτροπές ε, ε Ήτρε και για να ακολουθηθεί μια κοινή προσέγγιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το θέμα. Προτείνω να εθετηθεί ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και προτείνω να υπάρξει ε, θεσμικός διάλογος με τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ούτω ώστε να υιοθετηθεί μια ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση, ευρωπαϊκός νόμος σε αυτό το τομέα και να εγκριθεί και τροποποίηση της ισχύουσης ε, νομοθεσίας η οποία δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που έφτιαξαν οι δύο προλαλήσαντες και πολλοί άλλοι που πήραν το λόγο και εκφράστηκαν. Εάν το κάνουμε αυτό θα ενθαρρύνουμε τεχνολογική πρόοδο και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους και αυτό θα μας βοηθήσει να διασκεδάσουμε και τις ανησυχίες των πολιτών μας. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την εκμετάλλευση αυτών των πηγών. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι χρειάζεται μια στρατηγική αξιολόγηση των συνεπειών για το περιβάλλον. Όχι μια απλή αξιολόγηση, διότι πρέπει να εξετάσουμε και τα σωρευτικά αποτελέσματα οι διαδικασίες αυτές είναι περιπλοκότατες και μόνο με στρατηγική αξιολόγηση συνεπιών για το περιβάλλον μπορεί να αντιμετωπιστούν. Χρειάζεται να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός νόμος, ευρωπαϊκή νομοθεσία, ούτω ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, πληρούνται οι σωστέ απαιτήσει που δεν επιβάλλονται από τι πολυεθνικέ, αλλά από, τους, ε, από την πανεπιστημιακή κοινότητα, του ακαδημαϊκού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν το κάνουμε αυτό, διαφορετικά θα είμαστε θύμα των συμφερόντων των πολυεθνικών εταιριών που δεν είναι πάντα φιλικές για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Ζημάσκη. Ο Ζημάσκη. Αυτή τη φορά έχω μια ερώτηση, λέει ο κ. Ζημάσκη. Σύμφωνα με τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, θεματοφύλακα του νομικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ακούσω το σχόλιο σας για το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε επίσημη δήλωσή της δηλώνει σαφέστατα ότι το κοινοτικό κεκτημένο, το ισχύον νομικό πλαίσιο, αν εφαρμοστεί σωστά στα κράτη-μέλη, καλύπτει πλήρως όλα τα προβλήματα σχετικά με την εξαγωγή, διερεύνηση και εκμετάλλευση του συστολιθικού αερίου, άρα δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε οτιδήποτε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, διότι ήδη παρέχονται οι αναγκαίες προδιαγραφές για αυτή τη συγκεκριμένη ε, βιομηχανική δραστηριότητα. Καλύπτεται αυτή η συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα νομικά. Ευχαριστώ. Wills. Λέγομαι Σαβίνε Βίλτς, είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είμαι από τη Γερμανία. Κάθε πρωτοβουλίες κατά της υδρορογμάτωσης θα ήθελα να τις ενθαρρύνω ιδίως αν γίνονται επί τόπου. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τις σοβαρά αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σήμερα παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα, ότι μολύνεται το κόσμο νερό στη Γερμανία. Το συζήτησα με τον οργανισμό του Ποσίμου Ήδατος και με την ομάδα των αριστερών στο Κοινοβούλιο. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς ε, και από ποια σημεία περνάει το πόσιμο νερό, ποιε είναι οι διαδρομέ του και ξέρετε πω ε, το πρόβλημα τη μόλυνση είναι διαμεθοριακό. Πώ είναι δυνατόν αυτή η διαδικασία υδρορογμάτωση να είναι συμβατή με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Υπάρχει απαγόρευση τη ε, επιδείνωση του νερού. Άκουσα ότι οι χημικέ ουσίε αυτέ μπαίνουν στο έδαφο και δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν μετά την υδρορογμάτωση. Ότι η διαδικασία αυτή όταν ε, ξανανεβαίνει το νερό κουβαλάει και μια σειρά από βαρέα μέταλλα. Και δεν είναι δυνατόν να μην έχει αυτό επιπτώσεις και στα ύδατα και στις επιφάνειες, στην επιφάνεια μετά ε, του εδάφους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις για την υδρορογμάτωση, διότι σε πολλές χώρες, αυτή τη στιγμή όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες με βάση το δίκαιο για τα ορυχεία γίνεται η υδρορογμάτωση, δεν ε, γίνεται μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ως ομάδα και με άλλους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θεωρούμε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ρύθμισης. Εγώ θα ήμουν υπέρ του να μην επιτρέπεται καθόλου η υδρορογμάτωση και να δούμε μετά επί τόπου πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κολάσκα έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, άκρος ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Ε, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το σχιστολιθικό αέριο είναι αέριο όπως όλα τα άλλα. Χωρίς να κάνουμε τη διάκριση συμβατικού και μη συμβατικού. Η μη συμβατική πτυχή ποια είναι, ότι εξάγεται με κάπως διαφορετικό τρόπο. Διότι όταν μιλάμε για συστολιθικό αέριο, μου δημιουργείται ξαφνικά η εντύπωση ότι μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, που θα πρέπει να ρυθμιστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο νομικά. Ότι είναι κάτι εντελώς νέο. Όμως, βεβαίως υπάρχουν πολλές πηγές για να εξαγάγουμε και να εκμεταλλευτούμε το αέριο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νομοθεσία, για τη συγκεκριμένη πηγή του αερίου, διότι δεν μιλάμε για διαφορετικά ορυκτά καύσιμα εδώ, όπως είναι το πετρέλαιο και τότε θα έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί η νομοθεσία με τον δεδειγμένο τρόπο για να καλύπτεται η άλλη πηγή. Αναφερόμενοι τώρα στα όσα μας είπε ο κύριος Μποστινάρου. Αναφέρθηκε στα μονοπόλια ο κύριος Μποστινάρου. Τα μονοπόλια που μας υποχρεώνουν να κάνουμε κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι τα μονοπόλια του αερίου δεν ενδιαφέρονται στην, ε, για τη διερεύνηση και εξόριξη του συστολιθικού αερίου διότι θα είναι επιβλαβές για τα ρωσικά μονοπόλια διότι η εξόριξη του συστολιθικού αερίου σημαίνει ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα πέσουν. Ε, άρα ε, δεν μας πιέζουν να κάνουμε κάτι τα μονοπόλια. Τα μονοπόλια δεν θέλουν να κάνουμε κάτι για το συστολιθικό αέριο. Δεν θέλουμε να ανακτήσουμε το συστολιθικό αέριο. Αυτό είναι ένα σχόλιο που είχα από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πάρω το λόγο για πολύ λίγο. Πρώτα απ' όλα θα σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών για τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου και αυτής της ακροάσεως που έχει σαν βασικό στόχο, ελπίζω, να ακουστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, να ακουστούν οι αναφέροντες, η συζήτηση όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο από το σχιστορίθο γίνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνει χώρα στην Επιτροπή Ήτρε και συζητήθηκε όλα. Υπάρχει πρόταση αυτές οι δύο επιτροπές να συνδεθούν σε εργασίες τους εν ώψη ενός ψηφίσματος. Εμείς στην Επιτροπή Αναφορών βρισκόμαστε τώρα για να ακούσουμε κυρίως τους Ευρωπαίους πολίτες, τους αναφέροντες. Εγώ, ε, μπαίνω στο νομικό θέμα όσον αφορά την ανεπάρκεια του κοινοτικού δικαίου σήμερα και έναντι αυτής της νέας τεχνολογίας και της νέας ενεργειακής πηγής λέγατε ότι δεν έχουμε ειδική νομοθεσία ανάλογα με τις ενεργειακές πηγές όπως με το πετρέλαιο κλπ. Ναι, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τελευταία καταστροφή την πετρελαϊκή επικαιρεώνουμε ε, όσον αφορά ε, τις, την ανάγκη για λήψη μέτρων πρόληψης όσον αφορά τα θέματα του πετρελαίου στη θάλασσα. Όσον αφορά το σχητολιθικό πετρέλαιο και το αέριο, είναι νέα τεχνολογία. Δεν έχει σχέση αν μιλάμε για συμβατική με συμβατική ενέργεια, γιατί το λέμε αυτό. Διότι η εξερεύνηση και εκμετάλλευση του συστολιθικού αερίου και πετρελαίου σήμερα γίνεται με έναν τρόπο που οδηγεί μέσω της χρήσης της τεχνολογίας στο αντίθετο το ερώτημα των αντικτύπων που δεν ετίθετο για την εκμετάλλευση τη συμβατική για το φυσικό αέριο, διότι γίνεται εις βάθος η εκμετάλλευση, διότι χρειάζονται, χρησιμοποιούνται χημικά, χημικές ουσίες που ρυθμίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσης, κυρίως από την οδηγία REACH, διότι έχουμε μια νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των υδάτων και εγώ ε, κα, καλώ την Πολωνία που καταδικάστηκε επανειλημμένα για μη σεβασμό της οδηγίας για πλαίσιο για τα ύδατα να τη σεβαστεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε την οδηγία, πλαίσιο για τα ύδατα και ανησυχούμε όσον αφορά τις αξιολογήσεις και τις μελέτες αντιχτύπου και είναι και πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό. Στα πλαίσια της αναθεώρησης των μελετών αντιχτύπου σε κλίμακα ευρωπαϊκή, ότι πρέπει να γίνει κάτι και ανακοινώθηκε, δεν επίσημο, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ και ένα χρόνο, Κάποιε μελέτε μα δείχνουν ότι νομικό σήμερα η διερεύνηση εκμετάλλευση των συστολιθικών αερίων και πετρελαίου δεν εντάσσονται στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο υπάρχει και χρειάζεται νέα ρύθμιση. Και ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργαζόταν νέα νομοθετική ρύθμιση. Άρα η συζήτηση που γίνεται, και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, ε, ε, δικαιολογείται απόλυτα και έχουμε ανεπάρκεια και ένα όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο σε σχέση με τη ενεργειακή πηγή, τις νέες ενεργειακές πηγές που απαιτούν ε, ειδικά μέτρα, ειδική κάλυψη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους. Ε, εδώ πρέπει να θέτουμε ερωτήσεις. Η συζήτηση θα γίνει στο τέλος. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Μπουρλάντ. Δεν έχω ερώτηση. Λυπάμαι που θα σα απογοητεύσω, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να βάλω και εγώ το πετραδάκι μου στο κτίριο αυτών που είναι κατά του σχιστού αερίου. Πολύ σύντομο λοιπόν θα είμαι. Συμφωνώ απόλυτα ότι από πλευρά περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είμαι στην Επιτροπή Απασχόλησης, ξέρω ότι η εκμετάλλευση του σχίστου αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε 600.000 καινούριε θέσεις εργασίας και βεβαίω και εμείς στην Ένωση θέλουμε θέσει εργασία, πολύ επίκαιρο και επίγον αλλά να καταστρέψουμε το περιβάλλον αυτών που θα δουλεύουν να τους δώσουμε δουλειά και να τους κάνουμε μετά να πεθάνουν σιγά σιγά δεν αξίζει τον κόπο είναι πολύ επίγον η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και ευτυχώς οι συμπολίτες μας ε, απευθύνονται σε μας και μας καλούν να κάνουμε κάτι για το θέμα αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μας προτείνει η Κομισιόν ε, νομοθετικές διεξόδους για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρόεδρος, ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. παρακολούθησα τη συζήτηση πολύ προσεκτικά και διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις ε, και πολύ έντονα συναισθήματα. Ε, πολύ χαχυποψία και ε, ερμηνεία προθέσεων γίνεται ένθεν κακήθεν. Οι αντίπαλοι του σχιστοαερίου θεωρούν ότι η υπέρμαχή του είναι βασικά ανδρίκελα της βιομηχανίας. Οι υπέρμαχοι του σχιστοαερίου θεωρούν ότι οι πολέμοι είναι υπέρ της Gazprom. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Με τέτοια αμοιβαία καχυποψία, με τέτοιους ισχυρισμού ε, ισχυρισμούς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όλοι ανησυχούμε για το περιβάλλον και θέλουμε να το προστατεύσουμε. Ωστόσο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει ότι θα απαγορεύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο βιομηχανικές δραστηριότητες. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αναλυτική ε, νομική ε, κάλυψη. Αλλά αν είναι υπερβολική αυτή η νομική ε, ε, οι απαγορευτικές οι νομικές διατάξεις, τότε θα καταστήσουμε ανέφικτη την ε, εξόριξη του σχίστου αερίου. Παρακαλώ, θέλω να κάνω έκκληση. Να είμαστε λιγότερο συναισθηματικοί και περισσότερο επί τη ουσία να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να επιτρέψουμε στου χώρε που θέλουν να εκμεταλλευτούν το σχιστό να μπορέσουν να το κάνουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Παρακαλώ να απαντήσετε. Δύο λεπτά, παρακαλώ. παρακαλώ. Μερικέ ερωτήσει έχουν ήδη απαντηθεί λέει η κυρία Για το πόσο είναι πλήρες το κοινωνικό κεκτημένο. Βεβαίως, το αναφέρει μια έκθεση που ανέλει μόνο την ενεργειακή πλευρά. Στις, στις άλλες μελέτες, στις άλλες μελέτες που διάβασα, αναφέρεται και συμφωνούν όλες οι άλλες σε αυτό, ότι υπάρχουν κενά στην τρέχουσα ενωσιακή νομοθεσία και εκπρόσωποι τύπου της Επιτροπής ε, επίσης ε, το τονίζουν αυτό. Εγώ δεν ε, έχω κάποια συμφέροντα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Απλώς ανέφερα τη βρήκε η οργάνωσή μου μιλιό. Απαντώντας τα ερωτήματα που μου θέσατε. Και με αντικειμενικό τρόπο θεωρώ ότι διαπίστωσα ότι υπάρχουν κενά. Απαγόρευση τώρα. Εκμετάλλευση του σχίστου αερίου. Υπάρχουν ε, δυνατότητες να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα προστάτευαν το περιβάλλον και από πλευράς ε, αερίων θερμοκηπίου. Πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ του οικονομικού ενδιαφέροντος και της ε, ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτά είναι βέβαια θέματα της πολιτικής. Από νομική πλευρά, πρέπει να υπάρξει επαρκής ρύθμιση και είναι δυνατή η επαρκής ρύθμιση που να προστατεύει το περιβάλλον. Η νομοθεσία για την εξόριξη και τους υδρογονάνθρακες καλύπτει μόνο ορισμένες πλευρές. Για παράδειγμα, η οδηγία περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αφορά την εξόριξη υδρογονανθράκων, αλλά με τον τρόπο που την αφορά δεν καλύπτει το σχιστό αέριο. Οι αδειοδοτήσεις λοιπόν για την εξόριξη υδρογων η οι απαιτησει για οικονομικες εγγυσει νομοθεσία κάθε πλευρά της παραγωγής ενέργειας. Για τα ορυχεία τα περισσότερα νομοθετήματα είναι εθνικά, μόνο μερικά ενωσιακά νομοθετήματα καλύπτουν κάποιες πλευρές της εξόριξης των ανθράκων και ορισμένα από αυτά τα νομοθετήματα δεν αρμόζουν για αυτή τη νέα μορφή εξόριξης και αερίου. Νομίζω ότι από νομική άποψη αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαγεστέρο, Να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Αναφορά που λάβαμε από τη Βουλγαρία ο Η αναφερόμενη κυρία Ντουσάνα Στράβκο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω προσωπικά και τη γραμματεία της ε, ΠΕΤΗ για την οργάνωση αυτού του εργαστηρίου. Πολύ επίκαιρο το θέμα, πιστεύω. Δεδομένων των εκθέσεων που έχουν υποβληθεί στις, εκθέσεις, στις επιτροπές και ΙΤΡΕ. Η Επιτροπή ΠΕΤΗ πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ένα είδος ε, διαμεσολαβητή. Διότι εσείς έχετε την ε, ε, δέσμευση και το καθήκον να υπερασπιστείτε τους πολίτες που αναφέρονται σε εσά. Ε, δεν θα μιλήσω αναλυτικά για την ρουμανική αναφορά, επειδή πρέπει να κερδίσουμε χρόνο και επειδή πολλά από τα θέματα που αναφέρονται στην αναφορά μας είναι παρόμοια με τα θέματα που περιέχονται και σε άλλες αναφορές. Είμαι βαθιά. πεισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που καλείται να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης. Με συγχωρείτε κύριε Σόρνικα, αλλά ε, δεν μου είναι δυνατόν να μην είμαι συναισθηματική. Φανταστείτε το χάρτη της Ευρώπης, των περιφερειών της Ευρώπης, με αναφέροντας από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γερμανία και άλλες αναφορές. Αν δείτε το χάρτη θα καταλάβετε πόσο διαδεδομένη είναι η ανησυχία για αυτή τη μορφή εξόριξης. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι εμπειρογνώμονες Είμαι υπέρ μιας πιο περιοριστικής νομοθεσίας, ωστόσο η Επιτροπή Αναφορών θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην προετοιμασία μιας έκθεσης, πιστεύω, που να υποβληθεί στην Ολομέλεια. Στην ε, έκθεση αυτή πρέπει να ε, τονίσουμε πόσοι αναφέροντες έχουν υπογράψει αναφορές, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βούλησή τους, την επιθυμία τους για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναλύσει τι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουμε. Διότι εάν σε όλες αυτές τις περιφέρειες θεωρούν οι πολίτες ότι μπορεί να υπάρξει ερήμωση του περιβάλλοντος τους και να λάβετε υπόψη σας ότι οι πολίτες σε αυτές τις ε, περιοχές είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά τονίζουν την περιβαλλοντική πλευρά του προβλήματος. Για τη Βουλγαρία δύο μόνο θέματα. Έχει υπάρξει ένα moratorium, αλλά υπάρχει μια ad hoc ε, κοινοβουλευτική επιτροπή που ασχολείται με το θέμα αυτό και υπάρχει κίνδυνο να αρθεί το moratorium. Άμεσο είναι ο κίνδυνος δεν ε, έχει λοιπόν απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τη Βουλγαρία. Ο κύριος Μποστινάρου ανέφερε ότι δεν υπάρχει επαρκής διάλογος με τα θεσμικά όργανα. Η αναφορά μας έχει υπογραφεί από 8.000 πολίτες. Και 50.000 περαιτέρω ε, πολίτες ζήτησαν να επισυναυθεί και η δική τους υπογραφή και θα στείλουν ε, και εκείνοι την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πολίτες θα ήθελαν να συνεχιστεί ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Επαφίεμαι λοιπόν στην Επιτροπή σας και λέω τα εξή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ομάδες πίεσης. Ξέρουμε ποιοι πιέζουν εκ μέρους των ε, μεγάλων εταιριών. Αλλά το λόμπι, η ομάδα πίεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είστε εσεί. Και σα εμπιστευόμαστε πλήρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και πρόεδρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Τερέζα Βόιντα έχει το λόγο για να παρουσιάσει μια αναφορά που λάβαμε από την Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ήρθα εδώ, ήρθα από την Πολωνία για να σας πω κάποια πράγματα για τον, το πώς επηρεάζει η, Ευρωπα... η πολωνική πολιτική σκηνή, ο πολιτικός κόσμος, το αέριο. Έχουμε το Βόριτς και το Κούτνο, δύο πόλεις, όπου εκεί δεν χρησιμοποιούμε το σχίστο αέριο. Έχουμε τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου. Ήδη ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις κοντά στο Κούτνο για το υπόγειο αυτό απόθεμα του φυσικού αερίου θα εγχυθεί διοξίδιο το άνθρακος υπόγεια, ούτως ώστε να εξαχθεί το φυσικό αέριο. Και αυτή η υπέροχη αγροτική περιοχή, πασίγνωστη στον κόσμο, που είναι γνωστή για τις παραδόσεις της, για τα folklore κλπ. κινδυνεύει. Και ήρθα εδώ να ζητήσω τη βοήθειά σας, διότι στην Πολωνία κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται. Ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας, από τον οποίο ζητήσαμε γραπτός να κάνει κάτι, για να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια, δεν μας απάντησε καν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς, ε, διότι ε, παρέπεψε την Επιτροπή μας στην Επιτροπή Αναφορών και είμαι ευγνώμων εκ μέρους εκατομμυρίων Πολωνών που φοβούνται να υπογράψουν την αναφορά μας, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο προς υπογραφή. Εγώ και οι αδελφοί μου συντάξαμε από κοινού αυτή την αναφορά. Υπήρξαν σεισμικές δονήσεις στο, στην περιοχή Διεκοπόλσκα στην Πολωνία και ξέρουμε ότι είναι αποτέλεσμα ε, της εξαγωγής ε, σχιστοαερίου οι Πολωνοί δεν θέλουν την εξόριξη αυτού του αερίου, δεν θέλουν τα δύο τρίτα της χώρας μας να ε, υποχρεωθούν να εξάγουν το φυσικό αέριο. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ε, σχιστό αέριο ή ε, οποιαδήποτε άλλη μορφή φυσικού αερίου. Δεν θέλουμε την εξαγωγή αυτού του αερίου. Ε, Ποιε θα είναι οι πιθανότητε να ζήσουμε με ασφάλεια και να διατηρήσουμε τον τρόπο διαβίωσή μα. Ευχαριστώ όλου του εμπειρογνώμονε που καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν απειλέ και ποιε είναι αυτέ οι απειλέ. Όλοι γνωρίζετε πόσο νερό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ε, της υδρορογμάτωσης. Φοβούμεθα ότι θα χάσουμε την πρόσβαση στο ασφαλές, στο καθαρό πόσιμο νερό και περί αυτού πρόκειται η οδηγία πλαίσιο ε, για τα ύδατα. Εγγυάται την πρόσβασή μας σε καθαρό, εύγευστο νερό. Εγώ κατάγομαι το Wovitz, που από το Μάιο δεν πίνεται το νερό της βρύσης, δεν χρησιμοποιούσα καν το νερό της βρύσης εκεί, ούτε στο λουτρό, διότι δεν είμαι σίγουρη για την ποιότητα του νερού. Ε, εδώ και 40 χρόνια ξεκίνησαν οι πρώτες γεωτρήσεις εκεί και δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μολυσμένο το νερό. Ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας για την περιοχή μου για τη χώρα μου, για την πατρίδα μου, την Πολωνία. Ήρθα μαζί με την αδελφή μου. Ε, είμαι ευγνώμων, είμαι θα ευγνώμων, ευγνώμονες προς την Επιτροπή Περι, Περιβάλλοντος και ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει το ταχύτερον ε, δυνατόν. Διότι ακόμα και η καλύτερη νομοθεσία δεν θα εγγυάται την ασφάλειά μας. Η αδελφή μου και εγώ παρακολουθούσαμε εκ του σύνεγγυς τις διάφορες νομικές αλλαγές που επήλθαν. Ε, κυρίες και κύριοι, ο νόμος εμπόδισε τα δραματικά ατυχήματα στο Μπετούφ, το ατύχημα στο Μπετούφ στην Πολωνία και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Ξέρουμε ότι ε, οι υγρά απόβλητα έχουν ξεχυλήσει ε, και έχουν διαχυθεί και δεν μας είπε κανείς τι, περίχε το, τι περίχαν τα υγρά απόβλητα και ξέρουμε ποιες είναι οι δραματικές συνέπειες του ατυχήματος. Ίσως μια τέτοια συναισθηματική παρουσίαση, ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην την βλέπουν με καλό μάτι, με προειδοποίησαν γι' αυτό, αλλά σας παρακαλώ έχετε τα αυτά υπόψη σας. Στην Πολωνία αισθανόμαστε ότι απειλούμεθα. και η απειλή που δημιουργείται από την εξαγωγή του αερίου από εταιρείε που δεν ε, έχουν υπόψη τους τα δικά μας συμφέροντα και η νέα νομοθεσία επίσης ε, λησμονεί και τα συμφέροντα και η νομοθεσία λησμονεί τα συμφέροντα μας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι δύο αναφορές που παρελήθησαν από την Πολωνία δεν είναι παρόντες οι αναφέροντες και οι δύο αναφορές εφιστούν την προσοχή μας επί του εξής. Η Πολωνία κινείται προς εντατική εκμετάλλευση του συστολιθικού αερίου που αυτό ίσως συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα υπό τη μορφή ρήπανση των υπογείων υδάτων με χημικές ουσίες και μεθάνιο και αναφέρει αναφορά ότι οι συνολικές εκπομπές του διοξιδίου του θα είναι πολύ μεγαλύτερε από την απαγόρευση καύση άνθρακα. Ζητάει αναφορά, με αναφορά στο άρθρο 194 παρέμβαση και απαγόρευση τη εξαγωγή ιστοριστικού αερίου που δεν θα δημιουργήσει μόνο καταστρεφικέ συνέπειε για το περιβάλλον και η μόλυνση αλλά και σοβαρέ απειλέ κατά τη ανθρώπινη υγεία και τη υγεία των ζώων. Κυρίω η δεύτερη αναφορά ζητά απαιτεί την άμεση πάυση γεωτρήσεων και την απόσυρση των πολωνικών και των ξένων εταιριών. Θα δώσω το λόγο τώρα στον πρώτο από τους δύο εμπειρογνώμονες που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ε, καλύτερα το όλο ζήτημα. Δόκτωρ Μισελ Λαμπέλ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθώ στις ε, αναφορές αυτές των πολιτών από τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Είναι τιμή μου που μου ζητείτε να το κάνω αυτό και ελπίζω να το έχω κάνει αυτό, να το κάνω υπεύθυνα και να βοηθήσω να καθησυχάσω ε, τις ανησυχίες τους και να καθησυχάσω και υψηλότερα πολιτικά επίπεδα. Βλέποντα ανησυχίε για το συστολιθικό αέριο στη Βουλγαρία και την Πολωνία, όταν εξέτασα το θέμα, προσπάθησα να καταλάβω όχι τόσο τι τεχνικέ πτυχέ που νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκαν σήμερα και λεπτομερέστατα, αλλά να αναφερθώ στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στι πολιτικέ. Τι χρειάζεται να γίνει, τι μπορεί να γίνει, ούτω ώστε να καλυφθούν οι ανησυχίε του μακροπρόθεσμα. Και αυτό ξεκίνησα να κάνω. Η μεθοδολογία που ακολούθησα ήταν εξή ε, βασίστηκα σε πρώτες έρευνες που έκανα πώς μπορούμε να περάσουμε σε οικονομία μετά την οικονομία του άνθρακα και ναι, ε, δημιούργησα ένα πλαίσιο για τους κινδύνους, εξετάζω τους διαφόρους κινδύνους που αναφέρονται, το πώς λειτουργούν οι εταιρείε, πώς κινούνται οι κυβερνήσεις και πώς μπορούμε να απομακρυνθούμε από το παρόν ενεργειακό σύστημα που έχουμε και μετά εξέτασα τις αναφορές, τις ανησυχίες που εξέφρασαν στην Πολωνία και την Βουλγαρία και ανεφαρμόσα τον λόγο πλαίσιο. Πολύ σύντομα λοιπόν θα αναφερθώ σε κάποιες μικρολεπτομέρειες πριν φτάσω στα πορίσματά μου. Δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Μου ζητήθηκε να είμαι συντομότατο, λακωνικότατο και θα το κάνω. Αλλά τα πορίσματα και οι αναλύσεις θα είναι online διαθέσιμα στην πλήρη έκθεση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το πώ οι κρατικοί θεσμοί κινούνται και πώ οι εταιρείε κινούνται και πώς προχωρούν τεχνολογικά. Ε, και αυτό αξιολόγησα στις διάφορες συνεντεύξεις που έκανα στην Πολωνία. Έκανα 16 τις συνεντεύξεις και πράγματι ρώτησα τον κόσμο που εμπλεκόταν στον τομέα του συντοτικού αερίου ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες, ε, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι αν προχωρούσαν σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι και ο ρόλος της κοινωνίας και αυτό είναι ο ρόλος των ανησυχιών που αναφέρονται στις αναφορές και πάνω σε αυτά βασίστηκα στις ερωτήσεις που υπέβαλα στους, ειδικού. Η κίνδυνη είναι πολύ σημαντική διότι αυτά που αναφέρονται, οι κίνδυνοι που αναφέρονται στις αναφορές είναι σημαντικοί, αλλά επίσης και οι κίνδυνοι μπορούν να μειωθούν από τη χρήση στοριστικού αερίου είναι σημαντικοί. Και τι έκανα. Κατηγοροποίησα τις ανησυχίες που εκφράζει αναφορές και προσπάθησα να ανέβω σε επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, πίσω θεσμικός ο θεσμικό ρόλο των θεσμών στην Πολωνία. Εξέτασα αυτό. Το πώ οι περιβαλλοντικέ και τεχνολογικές ανησυχίε παίζουν ρόλο, οι οικονομικές επίσης ανησυχίες παίζουν ρόλο και να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να εξαχθεί το συστολιθικό αέριο ή όχι. Στην Πολωνία, πολύ σύντομα το λέω, μόνο 27 ε, Γεωτρήσεις έχουν γίνει, αναμένονται περισσότερες προς το τέλος του χρόνου, οπότε είμαστε ακόμα σε διερευνητική περίοδο στην Πολωνία και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη όταν εξετάζουμε τους κινδύνους και την, μελέτη, την περίοδο μελέτης που απαιτείται για την όλη διαδικασία. Ε, και εδώ βλέπουμε ένα χάρτη της Πολωνίας και που γενικά βρίσκεται σε αυτή τη φάση τη χρονική στο σχιστολιτικό αέριο. Είπαν ότι θέλουν 150 ε, δοκιμαστικά φρεάτια να δημιουργηθούν για να έχουν καλύτερη ιδέα για το εικόνα για το που είναι το συστηματικό αέριο. Η μεθοδολογία που ακολούθησα, 16 συνεντεύξεις έκανα και σε μεγάλη διάσκεψη πήγα που ήταν υπέρ του συστοριστικού αερίου, κυρίως ήταν υπουργοί της κυβερνήσεως παρόντες και κατάλαβα βέβαια ποια ήταν η άποψή τους. αυτό είναι το ενεργειακό μείγμα της Πολωνίας, άνθρακα, 90% του ηλεκτρισμού που παράγεται στη χώρα είναι από άνθρακα. Και βασικά όταν μιλάμε συστολιθικό αέριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε και για το ρόλο του άνθρακα στην Πολωνία. Λοιπόν, κάποια από τα βασικά πορίσματά μου είναι τα εξή. Είναι σχεδόν κρατικό πρόγραμμα και οι αναφέροντες στην Πολωνία θα συμφωνούν με αυτό. Πέντε διαφορετικά υπουργεία έχουν εμπλακεί στην διερεύνηση του θέματος του αερίου και την εκμετάλλευση αυτού και αυτό είναι σημαντικό διότι ε, κάνουμε ισολογισμό μακροπρόθεσμα. Πρέπει να δούμε κατά πόσο αν προχωρήσει το όλο θέμα πώς θα πει την νομοθεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ε, πώς θα κινηθούν οι εταιρείε όσον αφορά την εξαγωγή του συστολιστικού αερίου, πώς ελέγχονται κλπ. Λοιπόν, αποκρόθεσμα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή πώς οι εταιρείε, οι κρατικές εταιρείε και οι ιδιωτικές εταιρείε και το κράτος συνεργάζονται. Ε, τι αλληλεπίδραση υπάρχει. Και θα πρέπει να δοθεί βέβαια και στην κοινωνία των πολιτών φωνή στι συζητήσει. Και πρέπει να δούμε και για τι είναι σημαντικό το συστατικό αέριο στην Πολωνία, διότι υπάρχουν μεγάλε ανησυχίε για τον ασφαλή φοδιασμό σε ενέργεια. Και οι τιμέ είναι μια ανησυχία, ένα μεγάλο θέμα οι τιμέ, τιμολόγηση. Και αυτό είναι σημαντικό όταν δούμε ποιο είναι ο ρόλο των εισαγωγών υγροποιημένο φυσικό αέριο, εισαγωγή αερίου από την Ρωσία και το πώ η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα ορόσχη του ελληνικού αερίου που παράγεται ντόπια στην Πολωνία είναι κάτι σημαντικό, σημαντικό παράγον, ο οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τις οικονομικές και χρηματοστατικές πτυχές ε, του ενεργειακού μείγματος που ε, χρησιμοποιείται στην ε, Πολωνία. Επίσης, μία από τις αναφορές αναφερόταν και στις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σύγκριση με τις εκπομπές του από τον άνθρακα, από την καύση άνθρακα στην έκθεση. Είναι πολύ πιο λεπτομερή όλα αυτά, αλλά το συστατικό φυσικό αέριο έχει αντίκτυπο μεγάλη στη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο εν συγκρίση με το παρόν μείγμα άνθρακα στην Πολωνία και μελλοντικό μείγμα άνθρακα. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί, να, είναι, να λαμβάνεται υπόψη τη συζήτηση. Τώρα, από την έποψη την περιβαλλοντική είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι και ένα τμήμα τη συζήτηση. Και εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση και οι εταιρείε να ασχοληθούν με τι ανησυχίε που υπάρχουν. Οι περιοχέ του Natura 2000 είναι πάρα πολύ σημαντικέ, αλλά συνεντεύξει που είχαμε αξιωματούχου τη κυβέρνηση και των εταιριών Όλοι τόνισαν τη μεγάλη σημασία των περιοχών αυτών. Και ένα από τα μειονεκτήματα του συστολιθικού αερίου στη ΣΥΠΑ και αντίδραση κυβερνήσεων εκεί είναι ότι δεν άκουσα στην αρχή τι ανησυχίε των πολιτών. Και οι εταιρείε και η κυβέρνηση δεν ήταν αρκετά δραστήριοι στην αρχή, σε αυτή τη φάση τη της Πολωνίας εδώ και οι εταιρείε και η κυβέρνηση μπορούν πιο δραστηριοποιημένοι να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να προστατευτούν οι περιοχέ του Natura 2000 και θα μπορέσουν να επεξεργαστούν διάφορε συμφωνίε, ώστε η κοινωνία εν γέννη να μπορεί να καταλάβει τι διάφορε δυναμικέ που υπάρχουν, τι διαφορετικέ τεχνολογίε που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εξαχθεί το σχιστολιθικό αέριο με έναν τρόπο που είναι ασφαλέ προ το περιβάλλον και αν τελικά υπάρξει συμφωνία τη χρησιμοποιούμενη ε, τεχνολογία. Και μετά γρήγορα πάω προ τη Βουλγαρία. Υπάρχει ένα μορατόριο εκεί και η ανάλυση μου διαφέρει λίγο εδώ. Βλέπουμε το φυσικό αέριο, το μείγμα φυσικό αέριο στη χώρα και θα πρέπει να πω ότι η έρευνα που έκανα για Πολωνία και Βουλγαρία αφορούσε, ήταν και πρόγραμμα του 7ου προγράμματος πλαισίου. Έκανα συνεντεύξεις, δεν μπορούσα έγκαιρα να τελειώσω συνεντεύξεις για να υποβάλω αυτή την έκθεση, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο θα ληφθούν υπόψη που και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, τις πιο διευρυμένες, θα, τις, τα έχουμε του χρόνου. Λοιπόν, υπάρχει πάγωμα μορατόριο στη Βουλγαρία και πρέπει να δούμε τις πηγές φυσικού αερίου και κατά πόσο η Βουλγαρία ενδιαφέρει, ενδιαφέρει το ισοσορυφικό αέριο. Ε, υπάρχουν μεγάλα αποθέματα εκεί και ίσω εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει μακροπρόθεσμα να δούμε τι μπορεί να γίνει, ποιος είναι ο αντίκτυπος, όπω εξετάσαμε και στην Πολωνία. Εάν η τιμή, αν εισάγεται συμβατικό φυσικό αέριο με, με αγωγό αερίου και το κόστο είναι πολύ πιο χαμηλό από την εξαγωγή συστολιθικού αερίου στη Βουλγαρία, δεν υπάρχει οικονομικό επιχείρημα και δεν θα εκμεταλλευτούν το συστολιθικό αέριο στην Βουλγαρία, επειδή θα είναι πιο ακριβό και υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία στη Βουλγαρία, 90-95% εξάρτηση τώρα. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλγαρία θα πρέπει να έχει ποικιλομορφία όσον αφορά τι ενεργειακέ πηγέ τη. Ελπίζω να βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια τα διάφορα προϊόντα που παρέθεσα. Να Ναμπούκο, έχουμε το South Stream, του αγωγού. Έχουμε τερματικού σταθμού για υγροποιημένο φυσικό αέριο που οικοδομούνται, μεγαλύτερη, καλύτερη διασύνδεση που θα πρέπει να έχει η Βουλγαρία με τη γύρω περιοχή, όλα αυτά οδηγούν σε ποικιλομορφία όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα σε φυσικό αέριο για τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι αν το αέριο μπορεί να ε, έρθει από άλλε χώρε με διαφορετικέ μεθόδου, τότε δεν είναι τόσο ελκυστικό οικονομικά το σχιστολιθικό αέριο. Ελπίζω λοιπόν σε αυτή τη σύνοψη τη συντομότατη, σα είπα, θα είναι online διαθέσιμη πλήρη έκθεση. Αναφέρθηκα στι διάφορε κατηγορίε των ανησυχιών των αναφερόντων, ρυθμιστικό πλαίσιο, πλαίσιο πολιτική και μακροπρόθεσμα πώ αυτέ οι ανησυχίε μπορούν να διασκεδαστούν. Συντομότατα έχω κάποιε συστάσει για επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώση, γενικότερο επίπεδο. Πρέπει να δούμε ποιο θα είναι αντίκτυπος ε, των εκπομπών, σύγκριση άνθρακα και σχιστολιτικού αερίου. Για την Πολωνία είναι σημαντικό. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και θα το κάνω στο μέλλον και να δούμε κατά πόσο οι ανανεώσιμε πηγέ ενεργεία εκτοπίζονται το συστολιτικό αέριο. Αυτό που διαισθάνομαι είναι ότι περισσότερο ο άνθρακα θα εκτοπίσει το συστατικό αέριο από ότι ε, οι ανανεώσιμε πηγέ. Ανέφερα λοιπόν το ρόλο που παίζει η κρατική διοίκηση και πώ υπάρχει επαφή και συνεργασία με τι εταιρείε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ειδωθεί μακροπρόθεσμα. Και αν δούμε και άλλου ρυθμιστικού τομείς όπω είναι η ρύθμιση του τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια, η σωστή ρυθμιστική κατάρτιση για το διοικητικό προσωπικό είναι κάτι απαραίτητο, όπω έχονται σε επαφή και συναντούνται με τι εταιρείε, ποιε είναι οι επαγγελματικέ του γνώσει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά Υπάρχει η πιο νέα τεχνολογία, πρόσφατη τεχνολογία για τις ενεργές εταιρείε. Ε, είμαι πολύ ρεαλιστή σε αυτό και πιστεύω θα προχωρήσει όσον αφορά το συστολιθικό Άριο Πολωνία. Ποιε είναι οι σωστέ διαδικασίε, οι σωστέ κοινωνικέ επαφέ και συνανοήσει και μηχανισμοί που μπορούν να δημιουργηθούν στην Πολωνία. Αυτό είναι το θέμα για να επιτραπεί στην κοινωνία να εκφράσει την άποψή τη και να συμβάλλει στη διαμόρφωση τη χρήση τεχνολογία, πού χρησιμοποιείται, πώ χρησιμοποιείται. Και δεν μπορούμε πραγματικά, και το τονίζω αυτό, όντα στι Βρυξέλλε. Εγώ ζω στις, στη Βουδαπέστη, αλλά ο ρόλο του ασφαλού εφοδιασμού σε ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει σε κάθε συζήτηση για το συντηρητικό αέριο να συζητείτε. Κυρίω για την Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικό. Μπορούμε να συζητούμε αυτό το θέμα εδώ στι Βρυξέλλε, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και όταν μιλάμε για ενεργειακή ποικιλομορφία μακροπρόθεσμα, ο ασφαλή εφοδιασμό ο ενεργειακό έχει σημασία και η ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία σε μια χώρα και θα αναφέρω και τι θέσει εργασία γιατί είναι σημαντικό. Αν τα συζητάμε όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν διάφορε πηγέ για το ενεργειακό μείγμα και η τιμολόγηση τη ενέργεια τη χώρα παίζει ρόλο. Αυτέ οι χώρε λοιπόν, μιλάω για την Πολωνία, οι πολίτε δεν βγάζουν τόσα πολλά λεφτά. Υπάρχει μεγάλη ενεργειακή φτώχεια εκεί. Θα πρέπει σε κάποιο επίπεδο να αντιμετωπιστεί. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ καθηγητά κύριε Λαμπέλ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον καθηγητή κύριο Στάνης Λαυνάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαι εδώ σήμερα. Είναι η δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα και πέρυσι όπου άκουσα μία συζήτηση στην ίδια ακριβώς αίθουσα που είμαστε και σήμερα. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που ξαναβρίσκομαι εδώ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μία από τις πλέον σοβαρές ανησυχίες που ετέθη εδώ είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Έλλειψη αξιόπιστων ακριβών στοιχείων για τις τεχνολογίες, για τους κινδύνους Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα και ενοφανή ε, ζητήματα και έννοιες. Πρέπει όμως να υιοθετήσουμε μια ορθολογική προσέγγιση, ιδίως από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν να προχωρήσω, θα ήθελα να σχολιάσω την πρώτη παρουσίαση, την παρουσίαση του κυρίου Altman. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να θέσω υπόψη σας, φοβούμαι. Κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, αναφέρθηκε στι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, εξέφρασε κάποιε επιφυλάξει σχετικά. Εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά καμία απολύτω περίπτωση που να δημιουργεί ανησυχία. Αναφέρθηκε 5%. Αυτό μπορεί κανείς να το βρει ε, σε όλες τις συμβατικές περιπτώσεις, αλλά τα συμβατικά κοιτάσματα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα έπρεπε να ανησυχούμε. Άρα, να, μία ακόμη ανακρίβεια για την επίπτωση και για τα 500 μέτρα. Ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Ντέρεμ ε, μας δείχνει ότι 300 είναι τα μέτρα. Η παρουσίαση επίσης ε, περιέλαμβανε και άλλες ανακρίβειες. Αργότερα θα αναφερθώ. Τώρα, θα ήθελα να αναφέρω κάτι σε σχέση με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν και σχετίζονται με τα γεωλογικά ρήγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η πίεση μειώνεται. Δηλαδή δεν ρέει εντός των ρηγμάτων το αέριο, αλλά στα ανοίγματα. Πάντοτε υπάρχει κίνδυνος όταν δεν σφραγιστεί το άνοιγμα καλά. Είναι ένα επιχείρημα που έχει ακουστεί, ακούστηκε και εδώ και είναι και σωστό. Μου φαίνεται όμως ότι οι εκτιμήσεις ε, κινδύνων πιο πολύ αφορούσαν το διοξίδιο του άνθρακα. Ο δεύτερος ομιλητής ο καθηγητής ε, κύριος Αναστασίου έκανε μια πολύ ωραία παρουσία και τον ευχαριστώ για αυτό. Οι αναφορέ τώρα από την Πολωνία αφορούν ζητήματα τα οποία σας έχω καταγράψει και τα βλέπετε στη διαφάνεια. Τα επιχειρήματα που εκθέτουν οι αναφέροντες μπορούν να συνοψιστούν σε ορισμένα βασικά πορίσματα τα οποία θα σας σχολιάσω. αμφότερες οι αναφορές, όσο επίσης και οι βουλγαρικές, για την περιοχή Νόβι Πάζα. Δεν ξέρω τώρα αν συζητείτε ακόμη η βουλγαρική περίπτωση, αλλά θα ήθελα εγώ να σχολιάσω όλες τις αναφορές και να πω ότι πρόκειται για ένα άκρο επίμαχο ζήτημα. Γεγονό που σημαίνει ότι ενδεχομένω να μην μπορέσουμε να δώσουμε ναι. απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν. Θέλω πάντως να πω ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο ζωφερή, δεν είναι τόσο μελανά τα χρώματα όσο τα περιέγραψαν ορισμένοι από τους αναφέροντες. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ιδίω ό,τι αφορά το έδαφος την αντίστροφη ροή του νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις εκπομπές στον αέρα, τον ε, κατεπίδοντα σχεδιασμό για την πολιτική προστασία και το καθεξής. Μια εφημερίδα από το 1993, εδώ βλέπετε ένα δημοσίευμα, μπορείτε να δείτε πότε πρωτοαναφέρθηκε η λέξη αέριο από σχιστόλιθο σε, κάποιους, ε, σε κάποιες ε, καμίνους στη φούρνο στη, στο Δυτικό Καναδά συγκεκριμένα. Άλλη εφημερίδα τώρα από το 83 και το 87 δύο από κόμματα. Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίμαχα ζητήματα. σε σχέση με τις περιοχές ε, που περιλαμβάνουν φυσικό αέριο. Έχουμε μελέτη στο MIT το 2011. Φυσικό αέριο είχαμε κάποια συμβάντα τα οποία μελετώνται, εξετάζονται από την έρευνα. 20 έχουν να κάνουν με, σχετική, με πιθανή μεταφορά, μετανάστευση και μόλυνση. Ας δούμε όμως κάποιες ράσονες περιπτώσεις. Κάτω-κάτω τις βλέπετε, ατμοσφαιρική ε, ρήπανση. Εκρήξεις. Αλλά είναι πολύ λίγα αυτά τα συμβάντα. Αν δει κανείς πόσες πολλές είναι οι γεωτρήσεις της Αυτά είναι τα στοιχεία 2006-2011. Επανέρχομαι στα συμβάντα αυτά. Πάντως δεν φαίνεται στη διαδικασία της συνδρομάτων σε καμία περίπτωση να έχουν ε, ανέβει τα υγρά, τα αερογματικά στο έδαφος και να έχουν επιμολύνει το υδροφόρο ορίζοντα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση θα πρέπει να παρακολουθούνται πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα ζητήματα. Είπαν κάποιοι για πυκνοκατοικημένες περιοχές, είπαν ότι απαιτείται πάρα πολύ χώρος για αυτές τις δραστηριότητες ε, γεωτρήσεων εξόρυξης, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα ουσιαστικά. Και στο υλικό που σας έχω προσκομίσει θα το διαπιστώσετε, θα το διαβάσετε. Σίγουρα έχουν υπάρξει πάρα πολλές ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Ε, έχει αλλάξει, έχει, η τεχνολογία έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος εκ τότε. με 20.000 τετραγωνικά μέτρα σε ένα φρεάτιο βλέπετε στη διαφάνεια. Ο συγγραφέα Κιν παρουσιάζει νέες προσεγγίσεις, νέες τεχνολογίες. Ούτε αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Υπάρχει βιβλιογραφία σχετική που μιλάει για κάθετη ε, διείσδυση. Βλέπετε στην ε, οθόνη τις σχετικές πληροφορίες γιατί μπορεί να ρέει το νερό τι χρειάζεται να γίνει. Ο καθηγητής Αναστάζιου, όπως και ο καθηγητής Σάλτμαν, μίλησαν για τις χημικές ουσίες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες λοιπόν, αλλά έχουμε και τη νέα τεχνολογία, την πράσινη χημεία. Υπάρχουν δημοσιεύσεις, εδώ βλέπετε διάφορα συγγράμματα στην ε, διαφάνεια. Μπορείτε να συμβουλευτείτε και πρέπει να έχετε υπόψη ότι είναι τελείως διαφορετικές οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα. Η πρώτη πραγματική όμως έκθεση για την υδρογμάτωση, να ανέφερε ο κύριος Σιμάνσκι, έγινε από το, το Πολωνικό στο Γεωλογικών Ερευνών. Και το Ίδρυμα πετρελαϊκού καυσίμου. Βλέπετε ποια περιοχή αναλύθηκε στο Webbing στην Πολωνία. Έχετε κάποιες πληροφορίες για το βάθος, 3,5 χιλιόμετρα, 4.000 μέτρα το συνολικό βάθος ε, με την οριζόντια τομή 1.000 μέτρα μήκος. Ποια είναι τα αποτελέσματα της ε, μελέτης. Εν γέννη θετικά ήταν τα ευρήματα. Δεν υπάρχει μείζον κίνδυνος για το νερό. Δεν υπάρχει κίνδυνος ρήπανσης. Τα υπόγεια ύδατα δεν επηρεάζονται, οι πηγές ε, ύδατος δεν επηρεάζονται. Κάποια στοιχεία βλέπετε τώρα εδώ για τον αέρα. έκθεση Weebing. Βλέπετε τις παραμέτρους. Η χορύπανση. 53 δεσιμπέλ. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η Τώρα Ας δούμε τα επίπεδα συγκέντρωσης. Δεν έχει αλλάξει στο έδαφος η συγκέντρωση. Βλέπετε τα σχετικά στοιχεία. Βλέπετε πώς παρουσιάζεται όλη η κατάσταση. Τώρα, έρχομαι στην τεχνική της ρογμάτωσης. Πώς λειτουργεί. Σεισμός, φύσμπι. Και βλέπετε στα Φίτζη το σεισμό, πώς και βλέπετε πώς επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν οι ρογματώσεις για την ε, σεισμογένεια των περιοχών. Ουσιαστικά πρόκειται για μικρούς μικροσυσμούς, μικροδονήσεις. Δεν υπάρχει μείζον κίνδυνος. Κάποιες παράμετρο σε σχέση με το νερό. Δεν υπάρχει αλλαγή προ και μετά. Να δείτε όμως ε, το νερό το οποίο ξανανεβαίνει σε επιφάνεια, ακολουθεί αντίστροφη ροή, και βλέπετε κάποιες αλλαγές, 4.000 έως 52.000 και μετά 16.000 επανέρχεται. Άρα βλέπετε ότι κάποιες παράμετροι εμφανίζουν υψηλότερες τιμέ, όχι όμως δραματικά υψηλότερε. Και είναι και προσωρινό το αποτέλεσμα. Έξω και δεν υπάρχει κίνδυνος, μη φοβάστε, δεν είναι σημαντικά αυτά τα επίπεδα. Εάν σας ενδιαφέρει η έκθεση, φυσικά και είναι διαθέσιμη όλη η έκθεση αυτή, δεν θέλω να ψέλθω σε μεγάλες λεπτομέρειες. Θα ήθελα να αναφέρω όμως και τα επιφανειακά υδατά. Όπως βλέπετε, όλες οι τιμές είναι φυσιολογικές. Δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι δεν ε, παρατηρείται σημαντική επιδείνωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να επισημάνω και να τονίσω. Είναι το σημαντικότερο. Έρχομαι στα υπόγεια ύδατα δεν βλέπουμε αλλαγή στην ποιότητα, όπως αυτή αναφέρεται. Ο κίνδυνος βέβαια υπάρχει και πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση. Δεν είναι όμως σοβαρός ο κίνδυνος, δεν είναι μεγάλος. Απλά πρέπει να το παρακολουθεί στενά. Εν κατακλείδη να πω πρέπει να απορριφθούν αυτές οι αναφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που σας υπενθύμισα ότι πρέπει να τελειώνετε. Να περάσουμε τώρα στην παρουσίαση της αναφοράς που λάβαμε από το Βασίλειο από την κυρία Ρόσμαρη Ρέχτερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όσοι έχετε την υπομονή να ακούσετε, ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τους απλούς ανθρώπους. Ήθελα να παρουσιαστώ ενώπιόν σας και να σας ζητήσω να υπάρξει μορατόριο σε αυτήν την ε, πρακτική μέχρι να υπάρξει σωστά διατυπωμένη και χρηματοδούμενη ρύθμιση. Και επειδή δεν ήξερα όλες τις νομικές επιπλοκές, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει νομοθεσία για αυτή τη διαδικασία. Τέτοια ε, νομοθεσία λοιπόν σε όλη την Ευρώπη ξέρω ότι στη χώρα μου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς ρυθμίσεις. Και η αντιμετώπιση του ζήτηματο αυτού γίνεται κάθε μέρα πιο επίγουσα διότι λόγω της σημερινή οικονομικής κατάστασης οι κυβερνήσεις που δεν έχουν επαρκή χρήματα ψάχνουν για περισσότερα εισοδήματα και μια εύκολη λύση στα προβλήματα ενεργειακής προμήθειας. Η κυβέρνησή μας, ενώ προηγουμένως ήταν επιφυλακτική έναντι του σχίστου αερίου, όρισε υπουργό στο Υπουργείο Ενέργειας, που είναι γνωστός για τον έντονο ενθουσιασμό του για το σχίστο αέριο, τον σκεπτικισμό του, σκεπτικισμό του για την ε, θέρμανση του πλανήτη και την αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις. Προς το παρόν, ε, αυτές οι ρυθμίσεις είναι θέμα της αρχής για την υγεία και την ασφάλεια, με βάση τους κανονισμούς που αφορούν τις υπεράκτιες γεωτρήσεις. Αλλά υπερακτίως δεν υπάρχουν άτομα, δεν υπάρχει γη, δεν υπάρχουν δρόμοι και σπίτια. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό με ενημέρωσαν ότι αυτή η αρχή για την υγεία και την ασφάλεια δεν έχουν ούτε τους αναγκαίους πόρους, ούτε την ε, πραγματογνωμοσύνη για να ρυθμίσουν την ε, εξερεύνηση για το σχίστο αέριο. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αυτού του οργανισμού δήλωσε δημοσίως Μα τι να επιθεωρήσουμε ή να ελέγξουμε. Οι γιώτρες είναι κυρίως κάτω από το έδαφος. Το μόνο μέρος του Ηνωμένου Βασίλειου όπου έχει γίνει γεωρογμάτωση είναι η κομιτεία του Λάγκασερ. Η εταιρεία, η Quadrilla που έκανε αυτή τη γεώτρηση για τα δύο χρόνια που είναι εκεί κυρίως ε, αυτορυθμίζεται. Ούτε μία φορά ο οργανισμός αυτός για την υγεία και την ασφάλεια δεν έχει πάει να κάνει κανέναν έλεγχο, για παράδειγμα τι ποσότητα νερού ξανανεβαίνει, κανένας έλεγχος των χημικών ουσιών που μπαίνουν στην υδρορογμάτωση. Έγιναν δύο μικρές ε, σεισμικές δονήσεις. Ήταν όμως αρκετά σοβαρές ούτως ώστε μία γεώτρηση να θυγεί και δεν ξέρουμε ακόμη ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της βλάβης. Από ό,τι έμαθα επίσης, τα ύδατα που ανεβαίνουν μπαίνουν στο κανάλι του Μάντσεστερ, από όπου περνάνε ε, μαούνες. Οι κάτοικοι του Λάγκαστρ είναι κατά αυτής της εξόρυξη χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ρύθμιση. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για αυτούς πιστεύω. Και για να κερδίσουμε τι, εισοδήματα για το Υπουργείο Οικονομικών, κέρδη για τις εταιρείε. Αυτά είναι τα μόνα κέρδη. Ενώ οι απώλειες είναι πολύ πραγματικός ο κίνδυνος για τα ύδατά μας. Για κάθε ε, φρεάτιο χρειαζόμαστε 5 έως 9 εκατομμύρια γαλόνια νερού. Ένα μικρό ποσοστό ξανανεβαίνει στην επιφάνεια ω τοξικό μείγμα γιατί περιέχει μόνο τα χημικά τη υδρορογμάτωση, αλλά επίση έχει μολυνθεί και από άλλα υλικά που βρίσκονται στου σχιστολιθικού ε, σχηματισμού. Μπορεί να είναι αρσενικό, ε, φυσιολογική ραδιενέργεια, βαρέα μέταλλα, βερίλιο και κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο τμήμα του νερού παραμένει βαθιά στο υπέδαφος και χάνεται για τον κύκλο του ύδατος μονίμως. Στον κόσμο μας έχουμε όλο και λιγότερα νερά. Μπορούμε να δεχθούμε τέτοιες απώλειες. Αν δεν υπάρξει επαρκής ρύθμιση, η σχιστολιθική εξόρυξη θα μειώσει την ποιότητα της ζωής μας, θα μολύνει τις κοινωνίες μας, θα θίξει την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας και θα θίξει και τα οικοσυστήματα και θα μας εμποδίσει επίσης από το να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα που χρειάζονται αμέσως για να προωθήσουμε την διατήρηση ενέργειας και τις βιώσιμες μορφές ενέργειας που είναι τόσο απαραίτητες για να αποφύγουμε την περαιτέρω κλιματική αλλαγή. Αυτό το μέλλον θέλουμε για την Ευρώπη. Πρέπει επιγόντως να δράσουμε. Χρειάζεται ένα μορατόριο συνολικά στην Ένωση όπως ξέρετε τα ύδατα και ο αέρας δεν σέβονται σύνορα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μορατόριο μέχρι στιγμής να υπάρξει σωστά χρηματοδοτημένο σύστημα ρύθμισης. Υπάρχουν αλλακτικές λύσεις στο αέριο, δεν υπάρχουν αλλακτικές λύσεις στο νερό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο κυρία Ρέχτερ. Τώρα ο κύριος Κέβιν Άντερσον που αντικαθιστά τον κύριο Τζον Μπρόντερικ. Παρακαλώ. On the issue, I'm sorry. I'm going to be focusing very specifically θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Όχι τόσο πολύ όσον αφορά την ε, παραγωγή και εκμετάλλευση σχίστου αερίου, αλλά από την καύση του σχίστου αερίου. Το πήραμε. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Και συγκεκριμένα θα αναφερθώ στις χώρες του παραρτήματος 1. Είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ε, κλιματικής αλλαγής διαχωρίζουμε τις χώρες σε χώρες παρατήματος 1 που είναι κυρίως οι βιομηχανικές, άρα και οι χώρες της Ένωσης και άλλες είναι, στο... είναι οι χώρες μη παρατήματο 1. Ποιο είναι το σημείο κλειδί που θέλω να αναφέρω. Το φυσικό αέριο, άρα και το σχίστο αέριο, δεν είναι χαμηλού άνθρακα. 75% του βάρους του φυσικού αερίου είναι ο άνθρακας και όταν το κάψουμε έχουμε διοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι λοιπόν χαμηλού, χαμηλής ε, ε, περιεκτικότητας σε άνθρακα. Λέτε ότι ίσως να είναι καλύτερο το φυσικό αέριο από τον άνθρακα. Φυσικά. Αυτό ισχύει εάν εξετάσουμε τον ε, άνθρακα που είναι μέσα στο έδαφος. Αν στη χώρα σας χρησιμοποιείτε σχιστολιτικό αέριο ή φυσικό αέριο και δεν χρησιμοποιείτε τον άνθρακα, τον οποίο όμως εξάγεται αλλού, για το κλίμα συνολικά αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αντικατάσταση. Ο άνθρακας να μείνει ανεξόρυκτος για να βελτιωθεί η κατάσταση του κλίματος. Εάν εξορυχθεί, το σχιστολιτικό αέριο είναι χειρότερο για το κλίμα. Σημαντικό σημείο αυτό. Το φυσικό αέριο δεν είναι χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα. Τώρα, ένα γενικότερο πλαίσιο. Θα χρησιμοποιήσω κάποιε παραθέσει από τον επικεφαλή του οικονομικού Τμήματο του Διεθνού Οργανισμού Ατομική Ενέργεια. Να καταλάβουμε τι γίνεται όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Θα αυξηθεί ε, η μέση θερμοκρασία μέχρι το 2040-2050 κατά 3,5-4 βαθμούς Κελσίου. Εκεί πηγαίνουμε. Θα είναι πολύ ριζική η αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. Έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο εκπομπών τώρα. Επίση, λέει ο επιστήμον αυτόν, αυτός ότι αν δούμε τις τάσεις αυτές θα μπορούσε ακόμη τον παρόντα αιώνα να αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 6 βαθμούς. Είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας που τα λέει αυτά. Θα είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις για τον πλανήτη μας. Δεν είναι λοιπόν ε, λίγο περισσότερη ζέστη. Το μέλλον μας είναι 4, 5 ή 6 βαθμοί. Εκεί πηγαίνουμε και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι δεν θα τον επιτύχουμε αυτό το στόχο. Έχουμε πέντε χρόνια για να αλλάξουμε το, ενεργητικό, το σύστημα ενέργειας ή θα αλλάξει από μόνο του. Όπως μου είπε ο συνάδελφος Μπρόντρικ που λείπει, βεβαίως έχουμε τώρα την χρυσή εποχή του φυσικού αερίου, αλλά δεν είναι χρυσή εποχή, δεν είναι χρυσός αιών για την ανθρωπότητα. Για τον πλανήτη καθόλου. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Εδώ έχετε τη συμφωνία πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το έχουμε υπογράψει. Η σταθεροποίηση των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα πρέπει να γίνει σε τέτοιο επίπεδο που να μην υπάρξει επικίνδυνη παρέμβαση στο κλίμα. Φυσικά, όλοι θέλουμε να μην υπάρχει επικίνδυνη παρέμβαση. Όλοι συμφωνούμε. Αλλά τι είναι επικίνδυνο, τι εννοούμε επικίνδυνο. Ευτυχώς ε, μπορεί να μας πούν οι πολιτικοί και η κοινωνία των πολιτών με βάση τη δική μας ενημέρωση τι είναι αποδεκτή κλιματική αλλαγή και τι είναι επικίνδυνη. Μια συνενετική θέση. Θα ήταν σωστό να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από δύο βαθμούς. Και πρέπει να αναλάβουμε δραστηριότητα ούτω ώστε ισοτήμως να προωθήσουμε και να επιτύχουμε αυτό το στόχο με τη βοήθεια της ε, επιστήμης. Και αυτό το κάναμε και στην Κοπενχάγη και στο Κανκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ε, παρόμοιε διατυπώσει στα κείμενά τη, όπω και το Ρωμένο Βασίλειο. Πρέπει να μην ξεπεράσουν την προ-βιομηχανική θερμοκρασία, οι θερμοκρασίε μα κατά πάνω από 2-3 βαθμού. Ωραία, ξέρουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο. Ορίσαμε τον κίνδυνο, συμφωνούμε ποιο είναι ο κίνδυνο, είτε μα αρέσει. Οι δημοκρατικέ μα κοινωνίε συμφώνησαν με αυτού του στόχου, η διεθνή κοινότητα συμφώνησε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να επιτύχουμε αυτού του στόχου. Πρέπει οι αθρηστικέ εκπομπέ, δηλαδή συνολικά οι εκπομπέ, διοξιδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων θερμοκηπίου πρέπει να μείνουν σε ένα επίπεδο που να μα δίνει υψηλή πιθανότητα να μην περάσουμε του δύο αυτού βαθμού αύξηση. Δηλαδή να έχουμε 90 με 99% πιθανότητα να μην ξεπεράσουμε αυτού του δύο βαθμού. Συμφωνούμε λοιπόν και με αυτό. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε υπερβολικές εκπομπές. Πρέπει λοιπόν οι συνολικές εκπομπές να είναι τέτοιες που να μην υπερβούμε τους δύο βαθμούς. Τι πρέπει να κάνουμε ως επιστήμονες, ως κοινό, για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το 2012 είναι ήδη πολύ αργά. Ας είμαστε ειλικρινείς η συνάντηση κορυφή στο Ρίου είναι το 1992 και από τότε καθόμαστε και κοιτάμε τι εκπομπέ να ανεβαίνουν χρόνο το χρόνο. Πάει. Ήδη υπάρχει πολύ ψηλή πιθανότητα ότι ε, η πιθανότητα 50% να επιτύχουμε το στόχο μας. Είναι σαν να λέμε ότι κάθε φορά που στον δρόμο έχω 50% πιθανότητα να με χτυπήσει αυτοκίνητο. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε τώρα όσον αφορά το κλίμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, ότι μπορούμε να σταματήσουμε την ε, αποδάσωση. Α υποθέσουμε ότι μπορούμε να κατεβάσουμε τις εκπομπές από την παραγωγή ε, τροφίμων στο 50%. Ας υποθέσουμε, τότε το ερώτημα για μένα και τους συναδέλφους μου στο κέντρο Τίνταλ, τι θα γίνει με τον ε, τομέα εκπομπών από την ενέργεια. Αυτός με ενδιαφέρει τώρα τι μας μένει να εκπέμψουμε ως φυσικό αέριο και σχίστο αέριο για να έχουμε μια 50% πιθανότητα να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς αύξηση που είναι επικίνδυνο. Τα μαθηματικά τώρα είναι μπλεγμένα. Υπάρχουν ε, πολλά επιστημονικά, ε, επιστημονικές εργασίες που τις έχουν ε, αποτιμήσει οι επιστήμονες. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε το μέγιστο των εκπομπών το 2020, αν μιλήσετε με Ινδούς και Κινέζους, θα σας πούνε δεν πρόκειται να γίνει στην Ινδία και την Κίνα πριν το 2030-2040, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνουν ε, στο ίδιο σημείο για πολύ καιρό. Είναι λοιπόν μεγάλη πρόκληση. Αλλά κοιτάξτε πώ είναι η καμπύλη τώρα. Κοιτάξτε την καμπύλη. Εδώ βλέπετε το διοξείδιο του άνθρακα ανά δισεκατομμύρια τόνοι. Γίγα τόνοι τους λέμε. Μέχρι το 2050. Είμαστε εδώ τώρα, συνεχίζουν να αυξάνονται βλέπετε ότι πέρυσι ανέβηκαν κατά περίπου 3%, την προηγούμενη χρονιά κατά 6%. Αυτό είναι υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τη βιομηχανική επανάσταση. Ενώ είναι λοιπόν μεγάλο θέμα στην πολιτική σκηνή η κλιματική αλλαγή, οι εκπομπέ αυξάνονται πολύ ταχύτερα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία μα. Εάν φτάσουμε στην μέγιστη τιμή το 2020 που είναι ήδη μεγάλη πρόκληση και μετά πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει η καμπύλη, εδώ κάτω από την καμπύλη βλέπετε, αυτό μετράει. Αυτό μετράει για να επιτύχουμε τους δύο βαθμούς μόνο. Να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς. Εντάξει. Εάν δεν κατέβει αρκετά γρήγορα η καμπύλη, υπάρχει μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερος κίνδυνος να πάμε στους 3 ή 4 βαθμούς. Για να υπάρχει ένας μικρός, μια μικρή πιθανότητα να επιτύχουμε το στόχο, θέλουμε μετά το 2020 η μειώση να είναι της τάξης του 10 έως 20% κάθε χρόνο για περίπου δύο δεκαετίε. Για να έχουμε μια μικρή πιθανότητα να μείνουμε στου δύο βαθμού αύξηση για την ενέργεια, όπου πρέπει να μπει και το σχιστολιθικό αέριο. Αν μπορείτε να δείτε εδώ τι λέω. Είναι ότι μέχρι το 2035-45 δεν μα μένει καθόλου χρόνο για τι εκπομπέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε παγίδευση και αποθήκευση. Μόνο αν είναι 100%. Και κανείς δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε 100% παγίδευση και ε, αποθήκευση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μόνο ανανεώσουμε τότε και πυρηνική. Μόνο αυτές θα μας βοηθήσουν. Για να έχουμε μια μικρή πιθανότητα να αποφύγουμε επικίνδυνη κλιματική αλλαγή. Για να καταλάβετε όσοι είμαστε στα πλούσια μέλη του κόσμου. Τι υπογράψαμε είναι ότι πρέπει να γίνει ισότιμα αυτό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι φτωχότεροι πρέπει να έχουν περισσότερο περιθώριο για να βελτιώσουν την οικονομία του, άρα περιθώρια για περισσότερε εκπομπέ. Και εμεί που είμαστε πιο πλούσιοι, λιγότερα. Τι θα σημαίνει για μας λοιπόν αυτό. Για να έχουμε μια μικρή πιθανότητα λέω για δύο βαθμού. 40% μείωση τα επόμενα τρία χρόνια. 40% και για τα τρένα και τα αυτοκίνητα και τα ψήλια και τα αεροπλάνα και τα πλοία. 40% και 70% μέχρι το 2020 και 90% συν δηλαδή να αποφεύγουμε πλήρως τον άνθρακα μέχρι το 2030 για να μας μείνει κάποιο περιθώριο για τα φτωχά μέρη του κόσμου να βοηθήσουν να αποφύγουμε. Αργήσαμε πάρα πολύ, δεν κάναμε τίποτα από το 92 και μετά, άρα τώρα πρέπει να δράσουμε. Αν βλέπετε τα στοιχεία. Γιατί είναι διαφορετικά τα πορίσματα αυτά από αυτά που ακούτε συνήθως. Πρώτο σχόλιο. Δύο βαθμοί δεν πρέπει να είναι ο στόχος μας το 2050. Αυτό μπορεί να μας αρέσει εμά. αλλά δεν αρέσει την επιστήμη. Το μόνο που αρέσει την επιστήμη είναι οι αθρηστικές εκπομπές. Αν ορίσουμε ισότιμα μεταξύ των χωρών παράρτημα 1 και μη παράρτημα 1, τότε το δικό μας τμήμα θα πρέπει να κάνει σοβαρότερες μειώσεις. Να λάβουμε υπόψη επίσης εκπομπές από την απερίμωση και τα τρόφιμα. Να θυμάστε επίσης ότι πρέπει να καταργήσουμε τον άνθρακα όχι μόνο στην παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά στην παραγωγή ενέργειας συνολικά. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην Ένωση στα επόμενα 10 χρόνια. Θα είχαμε 20 ή 30 αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά δεν το κάναμε. Το φυσικό αέριο δεν είναι συμβατό με μια επιστημονική εκτίμηση για το πώς θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Αν θέλετε μη επιστημονική προσέγγιση, συνεχίστε ακόμη και αν υπάρξει παγίδευση και αποθήκευση του άνθρακα, θα πρέπει να μπορούμε να παγιδεύσουμε και να αποθηκεύσουμε όλο περίπου τον άνθρακα. Και κανεί δεν λέει αυτή τη στιγμή ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Άλλο σημαντικό. Οι προτεραιότητε τη έρευνα πρέπει να είναι τεχνολογίε χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα. Άρα όχι αέριο. Τελικό συμπέρασμα. Για τις χώρες που δεν είναι στο παράρτημα 1 μπορεί να υπάρχει μια μικρή δυνατότητα χρήσης του σχιστολιθικού αερίου για να μειώσουν τον άνθρακα, εφόσον όλες οι άλλες αλλαγέ γίνουν σωστά, αλλά θα πρέπει να βρουν τρόπους να παγιδεύσουν όλο τον άνθρακα και επίση να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο να μην χρησιμοποιούν άνθρακα. Για μας το σχιστό αέριο δεν είναι συμβατό ακόμη και με μια νερωμένη εκδοχή των ε, υποχρεώσεών μας, ακόμη και αν έχουμε αποθήκευση και παγίδευση. Εάν θέλουμε να σεβαστούμε λοιπόν τις δεσμεύσεις μας, δεν πρέπει να καίμε το σχιστό αέριο. Αν δεν θέλουμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, μπορούμε να το κάψουμε. Αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να υπάρξει ταχεία μείωση της ζήτησης για ενέργεια. Και πρέπει να περάσουμε σε ενεργειακά συστήματα πολύ χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία, ο καθηγητής Μάικλ Στίβενσον. I got up at four o'clock this morning, so... Ξύπνησα στις 4 το πρωί, οπότε σας υπόσχομαι ότι ένα δεκάλεπτο χρειαστώ το πολύ. Να εισάγω την ε, όλη έρευνα που έγινε στη Βρετανία, τη γεωλογική. Ανήκουμε στη Βρετανική κυβέρνηση. Είμαστε ανεξάρτητος φορέας, οργανισμός, δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά του σχιστολιθικού αερίου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε επιστημονικά στοιχεία στην κυβέρνηση και στους πολίτες, ώστε να αποφασίσουν αν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε ή όχι. Το κάνουμε με ισότιμο ουδέτερο τρόπο αυτό. Αυτό που μου ζητήθηκε ήταν να σας δώσω συνοπτικά μια εικόνα της κατάστασης του Ηνωμένο Βασίλειο για το σχιστολιθικό αέριο με σύντομη περίληψη και αυτά που θα πω θα αναφερθούν και στα στοιχεία που έθιξε ο Βρετανός αναφέρον. Ο τίτλος μου «Πόσο φυσικό αέριο και πόσο ασφαλές να εξαχθεί». Ένα από τα πράγματα που λείπει πραγματικά από τη συζήτηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε πόσο φυσικό αέριο υπάρχει και αυτό είναι τόσο σημαντικό διότι αξίζει. Αξίζει να το συζητάμε στο θέμα. Αξίζει να επενδύσουν οι επενδυτές Αξίζει να σκεφτόμαστε κινδύνους και ρυθμίσεις εάν δεν μπορεί να συμβεί κάτι δεν υπάρχει αρκετό αέριο. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πόσο ασφαλέ είναι να εξαχθεί. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι ε, σύμφωνα με κάποιες δημοσιευμένες πληροφορίες και άλλες πληροφορίες και τι μπορεί να κάνει η επιστήμη για να γίνουν κατανοητοί κίνδυνοι. Δεν θα μπω στον τομέα που καλύπτει ο Κέβιν που είναι πάνω από το έδαφος αν θέλετε, είναι το ίχνος άνθρακα του συστολιθικού ε, αερίου. Είμαι ένας προσγεωλόγος οπότε θα μείνω κάτω από το έδαφος. Πόσο φυσικό αέριο υπάρχει. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις και σύγχυση. Γιατί, διότι διάφορες έννοιες είναι συγκεχημένες. Ε, λίγη υπομονή ζητώ. Υπάρχουν στοιχεία για πόρους, για διαθέσιμα, και από θέματα, διαφορετικά στοιχεία και αναμειγνύονται από το τύπο και από εκείνου που ακούν τι πληροφορίε. Δεν κατανοούν τη διαφορά που υπάρχει και είναι εντελώ διαφορετικά τα στοιχεία. Πόροι. Αυτό το στοιχείο δείχνει πόσο φυσικό αέριο υπάρχει κάτω από το έδαφος. Το απόθεμα είναι τι μπορεί να καταφέρει να βγάλεις, ε, να λάβεις υπόψη τι οικονομικέ παραμέτρου ε, η άλλου παράγοντε, ποια ειναι η αποψη του κοινού Φερρυπίν για το αέριο. Υπάρχουν εντελώ διαφορετικά στοιχεία. Και ο παράγων ανάπτυξη, ο συντελεστή ε, ή ε, συνδέει τα δύο. Το ποσοστό του φυσικού αερίου που μπορεί να εξαγάγει από το υπέδαφο. Στη Βρετανία είχαμε ε, κάποιες εφημερίδες που δημοσίευαν στοιχεία ε, πόρων όταν εννοούσαν αποθέματα επεκράτησε πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση και καταναλωτές είναι μπερδεμένοι και το κοινό είναι μπερδεμένο, δεν καταλαβαίνει πόσο φυσικό αέριο υπάρχει, δεν ξέρει πόσο θα έπρεπε να ανησυχεί. Ας δούμε κάποιες βρετανικές εκτιμήσεις για να δείτε τα επίπεδα της σύγχυσης. Το BGS, η οργάνωσή μου, έκανε έναν υπολογισμό κατά προσέγγιση αποθεμάτων. Πόσο αέριο θα μπορούσε να βγάλει κανείς από το υπέδαφος. Για το 2010 ήταν ε, περίπου 5 ε, TCF 1,5, 5,3 μάλλον. Αν δείτε όμως μετά τους πόρους είναι πολύ μικρό. Οπότε αυτομάτως ήρθαν στο BGS και μας είπαν γιατί υποτιμάτε. Ε, δεν το κάναμε αυτό. Ήταν διότι εξετάσαμε συγκεκριμένο στοιχείο. Λοιπόν, η Advanced Resources, ένα άλλο φορέας που έκανε παρόμοιο υπολογισμού, είπε 97 TCF φυσικού αερίου. Αυτό αφορά τα αποθέματα Κίκος 20 TCF ανακτήσιμες πηγές, ανακτήσιμους πόρους το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε δηλαδή 5,3 και 20 συγκρίσιμα στοιχεία, τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Δεν είναι διότι οι γεωλόγοι είναι ανόητοι, είναι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς υπολογισμούς και εκτιμήσει για τα αποθέματα, μόνο μέσω ε, γεωτρήσεων ε, μπορείς να το κάνεις. Και όσο πιο πολλά γεωτρήσεις έχει τόσο πιο πολλά η ε, Κοντρίλερ κάνει συγκροτήσει στο Λάνκασερ. 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η άδειά τους και έχουν 100 ε, TCF ε, για υπολογισμό πόρων και όχι αποθεμάτων. Η IGAS, άλλη εταιρεία, εκτιμά άλλο στοιχείο. Αναμειγνύονται τα, οι διάφορες μονάδες, οι διάφορες εκτιμήσεις και έτσι επικρατεί η σύγχυση. Και ένα άλλο στοιχείο που οι εταιρείε τείνουν να λένε ότι έχουμε μεγάλα αποθέμα, μεγάλες ε, πόρους για το συστολιθικό. Η Eden Energy έχει άλλο στοιχείο, η Dart Energy άλλο στοιχείο. Οπότε υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις, ποικιλομορφία στοιχείων. Αυτό μπορώ να ανακοινώσω ότι η BGS κάνει αυτό που ελπίζουμε ότι είναι αυστηρή και διαφανής εκτίμηση των αποθεμάτων για το ε, τμήμα Διδιεύθυνση Ενέργεια και Αλλαγή Κλίματο και ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε τα απορίσματα του έτου. Το άλλο ερώτημα. Πόσο ασφαλή είναι η εξαγωγή του αερίου. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα και μελέτε. Ευτυχώ κάτι έγινε. έγινε. Πριν από δύο-τρία χρόνια δεν υπήρχαν στοιχεία και συγγράμματα στον αφορά την ασφάλεια. Και δεν υπήρχαν έγγραφα που ελεγχόταν από μοτίμως ε, ερευνητές. Ε, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Βέβαια δεν υπάρχει έλεγχος για όλα τα έγγραφα από τους ομότιμους. Λοιπόν, ποιοι είναι οι κίνδυνες, παραθέτουμε εδώ. Ε, μπορείτε να δείτε εδώ συνοψίζουμε τίποτα διαβάστε τα άθρα, στον τύπο κλπ. Σεισμοί, ακαιρεότητα των πηγαδιών, μόλις υπογείων εδάτων, αδιενέργεια, μεταφορά εξοπλισμών και απόβλητα, ε, εκπομπές στην ατμοσφαίρα, θόρυβος, μεγάλα ποσά, μεγάλες ποσότητες ύδατος χρησιμοποιούνται για την ε, υδρορυγμάτωση. Δεν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ε, διότι θα χρειαστούν ώρες να το κάνω. Θα μιλήσω για τους σεισμούς και μόνο τώρα. Ε, οι σεισμοί είναι το μόνο πραγματικό πρόβλημα που είχαμε στο συντολιθικό αέριο μέχρι τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δόθηκε μεγάλη προσοχή από τα ΜΜΕ. Δύο σεισμοί ικανού μεγέθους, ένα σεισμός ήταν 2,3, αισθητός από πάνω από 50 ανθρώπους. Αν θέλετε να δείτε τι έγινε του σεισμούς, βλέπετε τα επίκεντρα στην ιστοσελίδα του BGS. Είναι ελεύθερες πληροφορίες διαθέσιμες. Εκεί βλέπετε το πράσινο και το κόκκινο αστέρι. Τι κάναμε στο BGS. Εντοπίσαμε τους σεισμούς, είδαμε όταν συνέβαιναν, που συνέβαιναν, είδαμε τα ίχνη των σεισμών, το σήμα από τους σεισμούς, συγκρίναμε και είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δύο σεισμοί να προκλήθηκαν από την ίδια δραστηριότητα, διότι η δραστηριότητα ε, συνέπεσε ακριβώς με την υδρορογμάτωση, ήταν 10 ώρες μετά τη μέγιστη πίεση και με μεγάλη βεβαιότητα, με εύλογη βεβαιότητα είπαμε ότι η υδρορογμάτωση ε, προξένησε σεισμούς. Ε, είναι μια ένδειξη σημαντική πως η επιστήμη μπορεί να μειώσει τις υπερβολές, τους υπερβολικούς σεισμούς για το σχιστολιθικό αέριο. Μπορούμε να πούμε ναι αυτό συνέβη εκεί, ο σεισμός προκλήθηκε από την υδρορογμάτωση. Ε, απευθύνουμε μια έκκληση για λογική, για ορθολογική προσέγγιση. Κάποιο ομιλητή είπε να είμαστε λογικοί και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι παράδειγμα πώ μπορεί να είναι κανεί λογικό. Ε, έγιναν ενδιαφέρουσε εργασίε όσον αφορά τους σεισμούς αυτούς. Η Royal Society, η Royal Academy of Engineering ξεπώνησε μία έκθεση για την εξόριξη ε, του συστατικού αερίου και την υδρορογμάτωση και κατέχει στο συμπεράσμα ότι μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί ασφαλώς από τη στιγμή που γίνεται η σωστή διαχείριση της ε, διαδικασίας και αναφέρθηκαν και στο, στους σεισμούς, θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό. Να πω παρεπιπτόντως ότι δεν ταιριάζει αυτό με την έκθεση που ετοίμασε η EA για κάποιες πτυχές. Δηλαδή ότι κίνδυνος από την Royal Society για τα τυχώματα των ε, πηγαδιών θεωρήθηκε αρκετά χαμηλός, ενώ άλλοι διατείνονται ότι είναι υψηλός. Υπάρχουν διαφορές ε, αντίληψη όσον αφορά τον υπολογισμό των κινδύνων. Δεύτερη έκθεση που είναι σημαντική καλύπτει ειδικά τους σεισμούς. Ήταν μια έκθεση τριών ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων που εξέτασαν διάφορες εκθέσεις που ανετέθησαν από την Κουαντρίλα. Και αυτές οι εκθέσεις αφορούσαν τους σεισμούς, γιατί συνέβησαν, γιατί συνέβησαν εκεί που συνέβησαν και πώς μπορεί κανείς να χειριστεί στο μέλλον α, σεισμούς. Και βασικά το συμπέρασμα της έκθεσης ήταν απλό. Πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να γίνουν μικρές προεγχύσεις, αρχικές εγχύσεις, πριν γίνει η βασική έγχυση, να γίνει μια βολιδοσκόπηση και σε πραγματικό χρόνο να ελέγχει κανείς και για την υδρογρογμάτωση, πώ προχωράει η υδρογρομάτωση μέσω μικροσυσμικής τεχνολογίας και να εξετάσει και μεγαλύτερε εκδηλώσει, γεγονότα σεισμικά μεγαλύτερης κλίμακας. Και αν είναι πάνω από 0,5 αυτό το γεγονός θα πρέπει να σταματήσει αμέσω την υδρορογμάτωση. Είναι ένα σύστημα σαν έλεγχο τη κυκλοφορία. 0,5 ανάβει κόκκινο. Αν φτάσει στο 0,5 μειώνει την πίεση, αφαιρεί το νερό και αφήνει να ερεμήσουν τα πράγματα. Ε, είναι εξαιρετικά προσεκτική αυτή η έκθεση. Κάποιες εταιρείε είπαν ότι είναι πολύ χαμηλό το όριο, ότι δεν θα μπορέσουν να το κρατήσουν ποτέ τόσο χαμηλά. Αλλά όσον αφορά την αποδοχή από το κοινό και να έχει εμπιστοσύνη το κοινό σε αυτά που κάνεις, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει σε πολύ χαμηλό προσεκτικό επίπεδο. 0,5 είναι το ενδεδειγμένο επίπεδο κατά την άποψή μου. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμα δεν έχει λάβει απόφαση κατά πόσο θα συνεχιστεί η υδρορογμάτωση. Στο BGS κάνουμε δύο σημαντικά πράγματα όσον αφορά το συστολιθικό αερίο. Το ανακοινώσαμε πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα κάνουμε έλεγχο για τα υπόγεια ύδατα, εξετάζουμε αν υπάρχει μεθάνιο στα υπόγεια ύδατα πριν γίνει η υδρορογμάτωση. Γιατί θα ρωτήσει κάποιο, απλούστατα. Αν ξέρουμε πόσο μεθάνιο υπάρχει στο υπόγειο νερό, στα υπόγεια ύδατα, υπάρχουν αρκετέ μεγάλε ποσότητε μεθανίου στα υπόγεια ύδατα στο ΕΒ. Αν ξέρει κανεί πόσο υπάρχει, αν κάποιο κάνει ένα λάθο και μεθάνιο μπει στα υπόγεια ύδατα, ξέρει ότι έγινε. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά προσεκτική και πολύτιμη αυτή η προσέγγιση επιστημονικός. Αυτό κάνουμε και σύντομα θα τελειώσουμε τις βορειοδυτικές ε, περιοχές, εκεί που ίσως τελικά πραγματοποιηθεί η υδρορογμάτωση και δεύτερον κάνουμε και χαρτογράφηση για ένταση στα πετρώματα, στρες, ε, βλέπουμε που ήδη υπάρχει ένταση στα πετρώματα. Δεν είναι ορατή, αλλά υπάρχει ένταση στα πετρώματα και δίνει ένα προσανατολισμό. Δεν θα πρέπει να κάνει υδρογμάτωση όπου υπάρχουν υψηλέ εντάσει στα πετρώματα, διότι το κάνει θα δημιουργηθεί και υπάρχει ρήγμα, υπάρχει πρόβλημα. Άρα και εδώ δημιουργούμε μια βάση αναφοράς αν θέλετε και είναι πολύ σημαντικό. Ετοιμάστε ε, γραμμές αναφοράς διότι ξέρεις πού έχουν κάνει λάθη εταιρείε αντί τη αυτή περίπτωση δεν υπάρχουν αποκλήσει. Το επόμενο που κάνουμε είναι ζητάμε στοιχεία για την αξιολόγηση του πώ επηρεάζει το συστηματικό αέριο την αγορά ενέργεια. Το BGS απάντησε τρει από τι ερωτήσει που ετέθησαν και άλλε εταιρείε και φορεί ε, ακολουθούν την κατεύθυνση και νομίζω ότι και ο Κέβιν απάντησε σε αυτέ τι ερωτήσει. Πορίσματα λοιπόν. Ένα σημαντικό πράγμα για τη συζήτηση είναι δεν ξέρουμε πόσο συστοριθικό αέριο υπάρχει. Ας γίνουμε πιο ρεαλιστές γι' αυτό πριν αρχίσουμε και ενθουσιαστούμε, να δούμε πόσο αέριο υπάρχει, επηρεάζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Γιατί δεν ξέρει κανεί αν θα έπρεπε να επενδύσει. Και αυτού που διαμορφώνουν την πολιτική του επηρεάζει. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να επενδύσουν πολλά χρήματα. Αν δεν υπάρχει ε, ιστορικό αέριο, το, το κάνουν. Συγχαίρεται, δημιουργείται σύγχυση στο κοινό επίση. Στη Βρετανία σεισμοί ήταν η βασική περιβαλλοντική ανησυχή. Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα μελέτες από πολύ αξιόπιστους φορείς που είπαν ότι μπορεί να τους χειριστεί τους σεισμούς μέσω του συστήματος αυτό που είπα ε, κόκκινου και πράσινου φωτό σαν είναι η κυκλοφορία. Για να σταματήσει του σεισμούς η BGS, ο οργανισμός μου ξεκίνησε ε, μελέτες για όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα και την ένταση στα πετρώματα, γιατί πρέπει να έχει κάποιε βάσει αναφορέ, να ξέρει αν εταιρεία έκανε κάποιο λάθο, και μια κοινή η ε, ειδική επιτροπή είναι σημαντική για την ε, Βρετανία και ο 14ος γύρος αδειοδότησης, όπου η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καλεί τις εταιρείε πετρελαίου και φυσικού αερίου να ζητήσουν άδειε για εκτάσεις για φυσικό αέριο και δεν ξέρουμε πόσο θα ενδιαφερθούν οι εταιρείε μέσω του δημοσιοποιηθεί αυτή, αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η ανακοίνωση. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ θα παρατηρήσατε ότι έχει αλλάξει η πρόεδρος. Υπάρχει δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις. Ο συνάδελφος Τέιλορ ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές που μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Είμαι εδώ για να στηρίξω την κυρία Ρέχτερ την αναφέρουσα από την νοτιοανατολική Αγγλία που ανήκει σε μία από τις πολλές ομάδες ε, της ε, νοτιοανατολικής ε, περιοχής που πραγματικά έχουν ξεσηκωθεί από την ανησυχία τους για τις δραστηριότητες υδρορογμάτων στην περιοχή. Τους έχουμε ακούσει διάφορα φιλεγόμενα και για την ίδια τη διαδικασία της υδρορογμάτωσης και ένα γενικό σχόλιο, την αναγνώριση ότι οι κανονισμοί που ισχύουν αυτή τη στιγμή δεν είναι οι κατάλληλοι ε, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκεκριμένα το επίπεδο στο οποίο οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις απαιτούνται. Είναι πάρα πολύ υψηλά αυτή τη στιγμή τα επίπεδα για τη μέση εγκατάσταση δρορογμάτωσης και αυτό ε, το έχουμε δει και στην περσινή έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και το έχουμε επισημάνει. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ενισχύει το αίτημα να υπάρξει ένας ενωσιακός κανονισμός και ρύθμος του ζητήματος είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη διαφοροποίηση ε, ανακράτος μέλος. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνησή του χθες μόλις χθες δημοσιοποίησαν την πρόθεσή τους να προσφέρουν ε, φορολογικά ε, πλεονεκτήματα ε, στις εταιρείε που εκμεταλλεύονται το αέριο από σχιστόλιθο. 22 μίλια όμως από τη διάρκεια της μάχης η Γαλλία απαγορεύει ουσιαστικά την υδρογμάτωση. Δεν μπορεί να έχουν και δύο δίκιο και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και όλα αυτά δεν κάνουν κάτι άλλο από το να υπογραμμίσουν την ανάγκη να ρυθμιστεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον να εξεταστεί ο αντίκτυπος ε, του σχιστολυθικού αερίου. Και γι' αυτό συμφωνώ με, το, με την κυρία Ρέχτερ και την ομάδα της για απαγόρευση μορατόριου ε, της δραστηριότητας αυτής μέχρι ότου υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα. Δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα παραπάνω πέρα από το κέντρο Τίνταλ και τις ε, ενδείξεις και τα στοιχεία που μας παρουσίασαν από πλευράς κλιματικής αλλαγής, ε, τι είναι πιο ασφαλές για το σχιστολιθικό αέριο, να παραμείνει εκεί που βρίσκεται, στο υπέδαφος. Υπάρχουν μόνο οικονομικά επιχειρήματα, υπάρχουν ε, διάφορες τέτοιες ε, αιτιολογίες που αναφέρονται, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Και νομίζω ότι η Ευρώπη έχει πλέον τη δυνατότητα να έχει τα ενία και να βοηθήσει τις χώρες να καταλάβουν τι διακυβεύεται με αυτά τα οποία ορισμένες χώρες επιδιώκουν να πράξουν. Θα παρακαλέσω λοιπόν να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές και δι συγκεκριμένη της κυρίας ε, Ρέχτερ και να προβούμε στις δέωσες εννοείς. Ευχαριστώ. Έχει περάσει πολύ ο χρόνος. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ, ήταν μάλλον δήλωση όχι ερώτηση. Ευχαριστούμε τους δύο μιλητές μας. Δεν αναγνώρισα κάποια ερώτηση που κάνατε, αλλά ήταν ευχαριστίες. Τους ευχαριστώ και εγώ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημέρης διάταξης. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν βλέπω. Όχι. Ωραία. Να περάσουμε στο θέμα της ημέρης διάταξης. Ευχαριστούμε πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά ε, έχουμε πίσει χρόνο. Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η κυρία Μαγδαλένα Σταζινέσκη. Σταζινέσκου. Παρακαλώ. Ε, πού είναι. Είναι παρούσα. Παρακαλώ, έχετε, έχετε το λόγο 5 λεπτά. Η κυρία Καρίνα Φόπελ είναι παρούσα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μα δώσετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. πρέπει να υπάρξει μια στοιχειοθετημένη και αντικειμενική συζήτηση για τους κινδύνους και τις δυνατότητες ε, που μας δίνει το συστολικό αέριο και εδώ και στα κράτη-μέλη. Η ανταλλαγή απόψεων, κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη συμβολή στη συζήτηση αυτή. Είναι μια νέα δραστηριότητα αυτή. Έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η υδρορογμάτωση στην κλίμακα και με την περιπλοκότητα που είναι, είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Και κάθε εβδομάδα μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο για αυτή τη δραστηριότητα. Οι περισσότερε αναφορέ που συζητήθηκαν σήμερα καλούν για ένα μορατόριο ή για απαγόρευση της δραστηριότητας ε, σε σχέση με το σχιστολιθικό αέριο. Και επίσης λέγεται ότι υπάρχουν κενά στην υπάρχουσα νομοθεσία. Μία πρόσφατη μελέτη που δεν έχει δημοσιευθεί του Ευρωβαρομέτρου καταδεικνύει το 74% των πολιτών θα ανησυχούσαν εάν στην περιοχή του υπήρχε εκμετάλλευση του αερίου. Αυτό δείχνει ότι οι ανησυχίε που εκφράστηκαν εδώ έχουν ευρεία απήχηση. Οι κίνδυνοι είναι πραγματική, κατά τη γνώμη μας. Οι φόβοι του πληθυσμού είναι πραγματικοί. Ο βαθμός στον οποίο οι φόβοι είναι αιτιολογημένοι είναι κάτι που πρέπει να εκτιμηθεί σοβαρά. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την συνθήκη, τα κράτη-μέλη καθορίζουν τι συνθήκε για την εκμετάλλευση των ενεργειακών του πόρων και αποφασίζουν εάν ή όχι θα επιτρέψουν την διερεύνηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην περιοχή τους μη συμβατικών μορφών φυσικού αερίου. Τα κρατημέλη λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν τα αναγκαία μέσα για συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία και ιδιαίτερα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία, Εάν υπάρχουν μέτρα που επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές των κρατών μελών για το ενεργειακό τους μείγμα, μπορούν να ληφθούν, αλλά χρειάζονται ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο των κρατών μελών. Εξετάσαμε την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για το σχίστο αέριο και η αρχική ανάλυση μας το 2011 θεωρεί ότι οι πρακτικές για το σχιστολυθικό αέριο καλύπτονται από την υπάρχουσα ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η περαιτέρω ενημέρωση ωστόσο θεωρήθηκε χρήσιμη για να ε, διευκρινίσουμε εάν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από την ισχύουσα νομοθεσία. Στα πλαίσια μιας ευρείας διαδικασίας συλλογής πληροφοριών παραγγείλαμε μια έκθεση για να αποτιμήσουμε τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και άλλες παρεμφερείς νομικές πλευρές. Η μελέτη αυτή υπάρχει στο ίντερνετ, δημοσιεύτηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Η μελέτη αυτή καταλήγει ότι υπάρχουν μια σειρά από περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και νομικές και κάποιες ανασφάλειες ε, ε, δικαίωση σχέση με το πώς θα εφαρμοστεί η, εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστεί η νομοθεσία. Μέχρι στιγμής αυτό απόκειται στην ερμηνεία των κρατών μελών, ε, όπως υπόθηκε πολλές φορές σήμερα, και αυτό βέβαια οδηγεί και σε διαφοροποιημένη μεταχείριση των διαφόρων project. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα συντονίζει εσωτερικά τι εργασίε τη με τι υπηρεσίε που, που ασχολούνται με την ενέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν ε, εντοπιστεί. Εξετάζουμε την ενδεχόμενη ανάγκη να υπάρξει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να έχει διάφορες ε, μορφές. Όλες οι διαφορετικές επιλογές ε, από τις υπιότερες μέχρι το να φτάσουμε σε νέα νομοθεσία είναι ανοιχτά. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε δεόντως. Τι επιπτώσεις επίσης θα είχε κάθε επιλογή και αυτό θα το αναλύσουμε. Και σε ό,τι αφορά το προγραμματισμό των εργασιών μας, θα θέλαμε εντός του επόμενου έτους, του 2013 δηλαδή, να έχουμε κάπου καταλήξει. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι εάν και εφόσον ένα κράτος μέλος θέλει να προχωρήσει με το συστολιθικό αέριο, θα μπορεί αυτό να το πράξει με ασφάλεια και κατά τρόπο ε, αποδεκτό περιβαλλοντικά. Και τα μέτρα προστασίας ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών κινδύνων. Και όλα αυτά να γίνουν το μέγιστο πνεύμα διαφάνειας. Ετέθησαν αρκετά ζητήματα εδώ και είναι ε, και υπό εξέταση και συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ αυτών, σημαντικέ πτυχέ είναι η προσεκτική επιλογή των ε, περιοχών, ε, ταυτοποίηση κινδύνων, παρακολούθηση συλλογή δεδομένων, να υπάρχει ακαιρεότητα του φρεατίου, διαχείριση των υδάτων, η αποκάλυψη των χημικών που χρησιμοποιούνται και το καθεξής. Επίσης, διατάξεις των διαφόρων ε, ενισχύ Και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Αλλά να έχουμε υπόψη μας και τις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ε, της επιλογής που θα κάνουμε. Δατόπιση ε, προς παραγωγή και χρήση ενέργειας πιο ενεργειακά αποδοτική και με λιγότερες εκπομπές άνθρακα είναι προτεραιότητα. Πρέπει να αξίσουμε την ενεργειακή απόδοση, το μερίδιο των ανώσιμων πηγών ενέργειας, να μειώσουμε τις εκπομπές στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ε, στόχοι που δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Ολοκληρώνω με τα λόγια αυτά. Σημειώσαμε βεβαίως τις ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ. Θα τις λάβουμε υπόψη μας και στο έργο που έχουμε να στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για λόγους ε, χρόνου προτείνω το εξής. Δεν κλείνει, δεν λύγει ακόμη η συνεδρίαση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα μέλη τώρα μπορούν να κάνουν μια σύντομη δήλωση, αλλά όχι πάνω από ένα λεπτό, γιατί πρέπει και αναφέρουσα στο τέλος να πάρει το λόγο. Αλλά πρώτα μέλη της Επιτροπής. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση αλλά δεν ε, θέλω το λόγο γι' αυτό. Έχω μια ερώτηση στην Κομισιόν. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στο ίντερνετ υπήρχε ένα βίντεο του εκπροσώπου της ε, Επιτροπής για το Περιβάλλον που είπε ότι η Επιτροπή εργαζόταν επί μιας νομοθετικής προτάσεως για να ε, ρυθμιστεί η εξερεύνηση και εκμετάλλευση του σχίστου αερίου. Περί πρόκειται. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Σύντομα παρακαλώ. Κοιτάξτε, ε, όπως εξήγησα, αναλύουμε τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την πολιτική και των δεχομένων μέτρων. μία απόφαση δεν ελήφθη μέχρι τώρα ε, όσον αφορά νομοθεσία που θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέφνερ. Με ένα λεπτό, καλά θα είμαι σύντομος παρόλα αυτά. Το πρόβλημα, χαίρομαι που η Κομισιόν κατέστησε σαφές ποια σημεία εξετάζει και προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί το πρόβλημα είναι ότι ενώ το σκέφτεται η Κομισιόν, το θέμα αυτό και η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Και δεν είναι μια τεχνολογία που το χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε κάποιο εργαλείο. Είναι τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για να σκάψουμε τη γη που έχει νερό, που φυτρώνουν τα φυτά μας, τρώνε τα ζώα μας. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν σεισμών. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι αντιμετωπίσιμη όλη αυτή η κίνδυνη. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα μορατόριο είναι αναγκαίο. Ούτω ώστε να γίνουν αυτές οι μελέτες που θέλετε από οικονομική, οικολογική, επιστημονική, νομική πλευρά και μετά να υπάρξει ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν να πούμε από τη μία ότι εμείς το σκεφτόμαστε ενώ από την άλλη οι κίνδυνοι μεγαλώνουν μέρα τη μέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να συμφωνήσουμε με την αναφέρουσα και να υπάρξει μορατόριο μέχρι στιγμής που θα έχουμε μια λύση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ, Βολάντ. Ε, μας δώσανε 10 λεπτά οι Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ εκπροσωπώ όλους τους φορείς στη Γαλλία, στην περιοχή Ile de France, αλλά και σε όλη τη Γαλλία που είναι κατά του σχιστό αερίου. Δεν θέλουμε αυτή τη μορφή ενέργειας. Θα συνεχίσουμε την εκστρατεία για να εμποδίσουμε με κάθε τρόπο την εκμετάλλευση του σχίστου αερίου γιατί είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα του μέλλοντος του πλανήτη μας όπως είπαν οι προλαλήσαντες, όπως είπαν και οι εμπειρογνώμονες όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται και τονίζουν ότι όπως δεν μπορούμε να περάσουμε το δρόμο με κλειστά τα μάτια, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την μορφή ενέργειας. Ο γαλλικός λαός θα το επαναλάβει όλο και δυνατότερα. Οπότε ως κοινοβούλιο αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία που σας δίνετε, νομοθετήστε θαραλέα. Γιατί αν το 2015 πρέπει να μειώσουμε, να έχουμε μειώσει κατά 40% τα αέρια θερμοκηπίου δεν μπορεί να γίνει με αυτή την πολιτική. Ίσως οι καταστροφές να προκύψουν πριν το 2015. Το σπίτι μας καίγεται και εμείς συζητάμε να λέμε να καλέσουμε την πυροσβεστική ή όχι. Σας παρακαλώ, είναι ουσιώδες. Mm. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για λόγους ε, δικαιοσύνης. Ο κύριος Πόλακ από την ε, Πολεμική Αντιπροσωπή. Ένα λεπτό παρακαλώ. Παρακαλώ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Δεν θα αναφερθώ σε περιβαλλοντικές εκθέσεις, διότι η πολωνική θέση είναι σαφής. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τις πολωνικές εκθέσεις όσον αφορά την υδρορογμάτωση. Ο καθηγητής Νάγκη και άλλοι εμπειρογνώμονες αναφέρθηκαν σε αυτήν. Είναι μια έκθεση που συντάχθηκε από την Εθνική το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών της Πολωνίας και σε αυτή την έκθεση αναφέρονται σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές συμπεριλαμβανομένων και των σεισμικών δραστηριοτήτων του θορύβου, ποιότητα του σφαιρικού αέρα, ύδατα, υπόγεια και επιφανειακά. Η υδρορογμάτωση δεν επηρέασε ε, το περιβάλλον δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και η ζωή των υδάτων δεν μείωσε τα επίπεδα, ε, η χρήση των υδάτων δεν μείωσε τα επίπεδα του διαθέσιμου νερού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος απάντησε απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που είχαν τεθεί. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ένα εκπρόσωπο από τη ρουμανική πλευρά, υπάρχει κανεί από πλευρά Ρουμανία. Όχι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Γιώργη Ντούτσαμ ε, λέγομαι και είμαι πρόεδρος της Εθνικ, του Εθνικής Υπηρεσίας για, τις, ε, για τους πόρους, τους ορυκτούς στη Ρουμανία. Ασχολούμαστε στην Ρουμανία με την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η έλλειψη επικοινωνίας και η έλλειψη πληροφοριών οδήγησαν στο να ζητηθεί απαγόρευση της χρήσης ορισμένων τεχνολογιών. Δεν πιστεύω ότι φτάσαμε σε μια στιγμή όπου μπορούμε να προτείνουμε περιορισμό όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιορισμό, επιτρέψτε μου να υποβάλω στην Επιτροπή, στη Γραμματεία της Επιτροπής σας, ένα έγγραφο που εμπεριέχει την άποψη του φορέα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που κρατήσατε το χρόνο ομιλίας. Αυτό ισχύει για όλους. Φυσικά μπορείτε γραπτώς να αποστείλετε στη γραμματεία μας και τώρα ε, η αναφέρουσα ένα λεπτό ε, παρακαλώ η καθεμία γιατί μετά θα πρέπει να σταματήσει η διερμηνία. Παρακαλώ λοιπόν πολύ σύντομα η καθεμία χωρίς μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας παρακαλέσω να μην ε, απορρίψετε την αναφορά μας γίνονται ορισμένε αναφορές ε, στα έγγραφα που έχουμε συγκεντρώσει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα έγγραφα. Πολυνικοί φορεί έχουν εκπονήσει αυτά τα έγγραφα. Τώρα το ερώτημα είναι. Είναι ένα πράσινο νησί, είναι μια όαση η Πολωνία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στην Πολωνία. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να πεθύνουμε στους Πολωνούς εμπειρογνώμονες. Σήμερα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την άποψη του πολωνικού λαού. Εσείς μπορείτε να καταλήξετε στα δικά σας συμπεράσματα αφού ακούσατε τους εμπειρογνώμονες, αλλά ακούστε και εμάς σας παρακαλούν πολύ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Πολωνίας το Σεπτέμβριο του 2011 μας ενημόρωσε λέγοντας ότι υπάρχουν πάνω από χιλιάδες ε, γεωτρήσεις ε, που θα γίνουν με υδρορογμάτωση. Δεν ξέρω τώρα για τα στοιχεία εδώ, δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μια επιστολή που στείλαμε στους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Άντων γράφει συγκεκριμένα, το οποίο παραπέμψε με αυτά που έλεγε, ε, το διαβάσετε και να δείτε και στο YouTube ένα βίντεο το οποίο δείχνει τους ε, κινδύνους ε, για, από την έκκληση μεθανίου στις ε, γεωτρήσεις. Σας παρακαλώ, σας κλιπαρώ, δράστε γρήγορα, πάρτε γρήγορα πρωτοβουλίες. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Σας παρακαλώ, δείτε το θέμα από την ηθική του σκοπιά αν θέλουμε να ζήσει, να παραμείνει η Ήπειρος ζωντανή και ο πλανήτης ολόκληρος, θέλουμε τη βοήθειά σας, γιατί κανείς δεν μας υποστηρίζει. Μεγάλο χειροκρότημα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας στηρίζουν, βλέπουμε, οι βουλευτές σας. Εμάς όμως, Πολωνούς, ποιος μας υποστηρίζει, μας αφήσανε μόνους μας το έλεος της μοίρας μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Προσέξτε όμως και θυμηθείτε αυτά που σας είπαμε. Σας δείξαμε επίσης ε, στοιχεία, σας φέραμε έγγραφα. Σας παρακαλούμε, μελετήστε τα, διαβάστε τα. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ. Ακούστε, ήρθα εγώ σήμερα εδώ, έχοντας ήδη εκ των προτέρων ε, πιστή ε, για πολύ λογικούς λόγους, για το ότι η εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής είναι άκρος εσφαλμένη πρακτική και όλα όσα άκουσα σήμερα επιβεβαιώνουν την άποψή Τι σύγχυση βλέπουμε να επικρατεί μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών απόψεων, τι έλλειψη κανονισμού παρατηρούμε, πόσο αδαείς είναι περισσότεροι ε, και από αυτούς που μάλιστα εφαρμόζουν όλα αυτά. Η διπλανή μου ε, είπε ότι εγώ ε, έχω προστασία, ε, αλλά μπορώ να σας πω ότι το μόνο που κάνουμε είναι σαν να χορεύουμε το χορό του Ζαλόγου, για πάνω να πέσουμε στον κρεμό. Σας παρακαλώ, πρέπει να υπάρξει απαγόρευση, να υπάρξει μορατόριο μέχρι ότου θεσπιστεί η νομοθεσία που θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξανά καλησπέρα. Με συγχωρείτε, χαίρομαι που έχει κάπως ε, αλλάξει η άποψη της Κομισιόν από τις 28 Φεβρουαρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, νομικές αβεβαιότητες και τους κινδύνους. Αλλά κυρίως επιμένω ότι μιλήσαμε πολύ σήμερα για την υδρορογμάτωση το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή καλό θα ήταν να διευρύνουν την ανάλυση τους για το θέμα αυτό και για τις άλλες μεθόδους που προκύπτουν η ε, ρογμάτωση με το διοξιδίο του άνθρακα, με το ήλιο, να λάβουμε υπόψη και τις άλλες ε, επιδράσεις που έχουν αυτές οι διαδικασίες ε, στο έδαφος, όπου υπάρχει μια γεώτρηση, σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τρία εκτάρια, οδική πρόσβαση, αγωγή, καμιόνια και δεν έχουμε καμία πείρα και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει διάβρωση των σωλήνων και να έχουν προβλήματα τις γεωτρήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τους ε, ε, συμμετέχοντες. 15 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Με μεγάλη, με μεγάλη γενοδορία παρακαλώ. 15 δευτερόλεπτα. να σας πω ότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλες αναφορές που θα λάβετε. Αναφορά Γερμανών πολιτών για το θέμα αυτό, Λουξεμβουργέζων, Βέλγων και εκ μέρους των ε, ψηφοφόρων μου θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση όχι μόνο να υπάρξει ψήφισμα, αλλά ίσω και μια γνωμοδότηση τη Επιτροπή Αναφορών, μια που υπάρχει τόσο ενδιαφέρον ε, στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να στείλουμε αυτή μας την άποψη στην, Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την Γραμματεία που, έκανε, που δέχτηκε το αίτημά μας. Πρόεδρος βεβαίω. βεβαίως. Στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Ως Επιτροπή Αναφορών νομίζω ότι ασχοληθήκαμε 3,5 ώρες με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ήταν σκόπιμο, όπως έδειξε και η συζήτηση, να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το θέμα αυτό. Διαπιστώσαμε ότι χρειάζονται νέες τεχνολογίες για αυτή την εξόρυξη, χρειαζόμαστε έρευνα, υπάρχουν κίνδυνοι. Επίσης έχουμε ανταγωνισμό με την πραγματικότητα που τρέχει και διαπιστώσαμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή ρύθμιση και νομοθετική ρύθμιση γιατί η Ήπειρός μας δεν μπορεί να διαχωριστεί. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να αναπτύξει αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προοπτική. Τέταρτο λοιπόν, σωστό και λογικό, να παραμείνουν ανοιχτές όλες οι αναφορές. Θα ασχοληθούμε πολύ έντονα με τα αιτήματά σας, διότι όσα αναφέρθηκαν είναι σημαντικά τόσο σημαντικά που εδώ μπορούμε να αρχιοθετήσουμε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ τους συμμετέχοντες, ευχαριστώ τους διερμηνείς που μας έδωσαν ένα τέταρτο και σας εύχομαι ευχάριστο βράδυ και καλό ταξίδι.